Καλημέρα σε όλους. Έχουμε μαζί μας και τους εισηγητές για διάφορα θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης, επομένως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το διαθέσιμο χρόνο. Θα ήθελα καταρχάς να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Θα ακούσατε ότι ε, ο κύριος Μπρόκ είναι ο εισηγητής για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Στις 28 ε, το απόγευμα θα γινόταν η συζήτηση, αλλά θα συζητήσουμε τελικά την έκθεση αυτή στις 4 ε, Μαΐου. Πρόκειται για μια μικρή λοιπόν αλλαγή που επιφέρουμε στη συζήτηση της έκθεσης αυτής. Μας ενημέρωσε η γραμματεία εγκαίρως και ήθελα να σας ενημερώσω στις αρχές της συνεδρίασής μας. Εγκρίνονται τα πρακτικά της 1ης Φεβρουαρίου και της 22ης και 23ης Μαρτίου και βέβαια εφόσον έχετε παρατηρήσει τροποποίηση και τα πρακτικά μπορείτε να μου το πείτε μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης. Θα ήθελα να καλωσορίσω στην ευρίασή μας τον κύριο Πιέρ Μορέλ, ο οποίος είναι ο ειδικό εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική Ασία και είναι εδώ σήμερα μαζί μας προκειμένου να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην Κυργιζία. Στις 20 Απριλίου η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Κάθριν Άστον μίλησε στην Ολομέλεια για τις εξελίξεις στην Κυργυζία. Ζητήθηκε από τον κύριο Μορέλ να πάει στην Κυργυζία μαζί με μία αποστολή των Ηνωμένων Εθνών και του ΟΑΣΕ προκειμένου να εξασφαλίσει μια πλήρη εκπροσώπηση της διεθνούς κοινότητας στη χώρα αυτή. Χαιρετίζω λοιπόν την αντιπροσωπεία και θα της δώσω το λόγο στην αρχή της συζήτησης. Δεν θέλω να κλέψω άλλο χρόνο από αυτήν την ενδιαφέρουσα συνάντηση. Δόκτωρα Μορέλ, σας δίνω το λόγο. Εσείς ε, θα αποφασίζετε πόσο χρόνο σας χρειάζεται, αλλά μην ξεπεράσετε τα 10-12 λεπτά για να μείνει χρόνο συζήτησης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση. Δεν είναι πρώτη φορά που έχω αυτήν τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την Κεντρική Ασία αλλά αυτή η φάση είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Και ελπίζω να ανταποκριθώ δηλαδή και στις προσδοκίες της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ακολουθήσω με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις οδηγίες σας και θα περιοριστώ σε μία παρουσίαση όσο δυνατόν πιο σύντομη και περιεκτική, έτσι ώστε να καλύψω τα κύρια ζητήματα, χωρίς απαραίτητα να επισέλθω στις λεπτομέρειες, γιατί αυτές μπορούμε να τις καλύψουμε τις ερωτήσεις. Είναι ένα ευρύτατο βέβαια θέμα και πρέπει να είμαστε ασφαλώς επιλεκτικοί. Κάθε μία από τις χώρες είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Θα το δούμε ιδιαίτερα με την Κυργισία αυτό, που είναι και το κύριο μας θέμα. Ξεκινώ λοιπόν με τα γεγονότα εκεί, στην Κυργισία προσπαθώντας να εξηγήσω το γιατί, το τι συνέβη. Διότι εξεπλάγησαν οι πάντες, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Δεύτερο θέμα, θα αναφερθώ στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πώς δηλαδή εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπόθεση αυτή, τι δεσμεύσει να λαμβάνει και επίσης παρατηρήσεις που είδαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ακούσαμε μάλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, από τη Λεδιάστον ε, και διάφορες παρατηρήσεις ε, που έχουν, διατυπωθεί, που έχουν εκφραστεί μετά τις ερωτήσεις για τη στρατηγική, για την Κεντρική Ασία. Είναι χρήσιμο λοιπόν νομίζω να κάνουμε και με κάποια σχόλια στην υπόθεση αυτή, αν δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη στρατηγική, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να είναι διαφορετική κτλ. Και θα προσπαθήσω και εδώ να απαντήσω στα ερωτήματα. Καταρχάς όμως το γιατί. Μια απλή απάντηση. Υπάρχουν και εσωτερικοί και εξωτερικοί λόγοι. Ή εσωτερικοί. Να ξεκινήσουμε αν θέλετε κι εσείς από τα πρόσφατα ε, γεγονότα. Η Κυργισία το 1992 προκύπτει ως ανεξάρτητη χώρα μετά την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια από τις δημοκρατίες αυτές που της έγινε ανεξάρτητη. Μια μικρή κάπως διαφορετική από τις υπόλοιπες, ε, όχι πολύ διαφορετική τέλος όχι πολύ ε, σημαντική δημοκρατία που έγινε ανεξάρτητη. Και με την υπόθεση που οδήγησε στο τέρμα την διακυβέρνηση του Αλκάιεφ, την επανάσταση του 2005, που πολύ γρήγορα αποεκλήθη η επανάσταση της Τουλίπας, και πολύ λίγο πολύ βλέπουμε να επαναλήφθηκε και τώρα, αλλά με διαφορετικούς Ε, ένα ειρηνικό δηλαδή κίνημα στο Μπίσκεκ που οδήγησε σε μια μεταφορά εξουσίας μετά από τις διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια, την κινητοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της αντιπολίτευσης, την αποχώρηση του Αλκάιεφ, του πρόεδρου Αλκάιεφ, ειρηνική επαναλαμβάνω, με διαπραγμάτευση χωρίς δηλαδή θύματα, πράγμα το οποίο δεν επαναληφθήκε τώρα δυστυχώς. Πάντως αυτή εκείνη, εκείνη η επανάσταση της Τουλίπας δείχνει πως υπάρχει βούληση του Κυργιστάν και του τμήματος της, ε, ενός τμήματος κοινωνίας, του λεγόμενου Ισλαμικού τμήματος, να ξεφύγει από τον εποτισμό λίγο πολύ. Γιατί... Απλουστεύω, αλλά αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν ένα κίνημα δημοκρατικό αντίδρασης, ειλικρινές και ξεκάθαρο μας στη χώρα, μια κοινωνία των πολιτών αρκετά ισχυρή, που έχει τη βούληση για την οργάνωση, για τις κινητοποιήσεις. Έχουμε διαρκή επαφή με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και στη συνέχεια αποσταθεροποίηση της εξουσίας θα έλεγα που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή κινητοποίηση που οδηγεί σε ε, βάλτο την κοινωνική ζωή, την, το κρατικό βίο, δηλαδή έχουμε τα διαρκή συλλαλητήρια. Από εκεί και πέρα ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει την διελκυστίνδα της δύναμης, προσπαθεί να κινητοποιήσει τους δικούς του ενάντια των υποστηρικτών του άλλου, υπάρχουν διαρκείς αντιπαραθέσεις στους δρόμους και ε, συγκρούσεις με τελική εκδήλωση την ανάληψη ε, της εξουσίας του ισχυρότερου σε αυτή την ε, πολλαπλή διελκυστίνδα που οδηγεί τη χώρα σε μία διολίσθηση προς το σύστημα των ε, φατριών θα έλεγα. Άρα έχουμε και αποσταθεροποίηση πολιτική και αγώνα για το ποιος θα εξασφαλίσει την εξουσία χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσον και φορέα και τελικά ε, κατάληψη του δημοκρατικού βίου από τις φατρίες, από τις μεγάλες οικογένειες. Αυτό έχει συμβεί τα τελευταία πέντε χρόνια και έτσι ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος που είχε ξεκινήσει με την ε, δυσφορία του λαού το 2004-2005 έναντι του Αλκίεφ και που τώρα μας έχει φέρει στο ερώτημα του πού πάει η Κυργυσία ποια είναι η κατάσταση από εδώ και μπρο, πώ θα ζήσει, πώ θα επιβιώσει. Και χωρίς να σα δίνω άλλες λεπτομέρειε, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τους οικονομικούς παράγοντες αυτής τη διολίστηση, διότι η οικονομική κρίση είχε τεράστιε επιπτώσει στο κράτος αυτό που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εμβάσματα των μεταναστών που έχει στη Ρωσία κυρίως και άρα εξαρτώνται πολύ από τα εμβάσματα. Όπω και το Τατζικιστάν εξάλλου που είναι το δεύτερο φτωχό κράτο κεντρική Ασία, συγκρινόμενο με τα πιο πλούσια κράτη που έχουν ε, ε, υδρογονάνθρακες και εκμεταλλεύονται. Τώρα, πολύ γρήγορα για να περάσω στην κυβέρνηση, είπα το, μίλησα για νεποτισμό, διαφθορά δηλαδή, για αποδιάρθρωση της εξουσίας σε εθνικό επίπεδο και σε όλο και μεγαλύτερη χειραγώγηση του πολιτικού συστήματος από τον Πρόεδρο και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης εξουσίας, μια αυταρχική δομή σιγά σιγά της εξουσίας ε, σε επίπεδο Προέδρου και οργάνωση γύρω από αυτόν κάποιων ολίγων. Ε, είχαμε αυθαίρετες συλλήψεις, είχαμε δολοφονίες, οι οποίες αντιδράσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα είχαμε και πολύ σημαντικές αυξήσεις τιμών σε αγαθά όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, που οδήγησαν τον κόσμο σε αντίδραση μερικές φορές και VA. Ο πρόεδρος προσπάθησε να αντιδράσει με το Κόλταϊ, με μια μεγάλη συνέλευση δηλαδή λαϊκή στην Επανάσταση του Λίπας, λέγοντας ότι πρέπει να αποδεσμευθούμε από τις παραδοσιακές μορφές της δημοκρατίας και η μορφή που αρμόζει προς τώρα στη χώρα μας, στην κεντρικό-ασιατική αυτή χώρα, είναι η συμβουλευτική λεγόμενη δημοκρατία. Για να σας εξηγήσω πόσο μακριά έχει πάει το πράγμα. Και στο Ταλά, στις 6 του μηνό, με την πρώτη μεγάλη διαδήλωση, αποφάσισε ο πρόεδρο να συλλάβει συλλήβδην όλου του αρχηγού αντιπολίτευση όλους. Εξού και κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης σε ένα τεράστιο συλλαλητήριο για να ε, διαδηλώσουν κατά της σύλληψης των αρχηγών της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, τις συνθήκες τις προκάλεσε η ίδια η πολιτική ε, αδεξιότητα, η κακή χειρισμή πολιτική και τελικά βέβαια καταλήξαμε με την τραγωδία στις 7 του μηνός ε, των πυροβολιστών μόν μπροστά στο προεδρικό μεγαρό με 87 νεκρούς για τους οποίους υπεύθυνο θεωρούμε τον πρόεδρο. Είναι η πρώτη φορά που ε, είχαμε τέτοιες τραγωδίες, ε, απώλειες ανθρώπινων ζώων, γιατί όπως είπα νωρίτερα ο Αλκάιεφ είχε αποχωρήσει ανέμακτα και η κατάσταση την οποία έχουμε τώρα μπροστά μα. Είναι νωρί βέβαια για να καταλήξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να κρίνουμε την κατάσταση συνολικά. Οι περισσότεροι λένε ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει αυτέ τι διολυστήσει. Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά σαφής η κατάσταση και δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εικόνε ε, παρεμβάσεων εκεί που δεν υπάρχουν πάντοτε. Απλώς θα ήθελα να πω ότι η Κυργισία που κανονικά δεν έχει καμία παρουσία στον ρωσικό τύπο, τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο διαπιστώσαμε ότι ε, καλυπτόταν με διάφορα άρθρα που έβαλαν κατά του καθεστώτος του Αλκίεφ, κατά της αναποτελεσματικότητάς του, κατά της έλλειψης δημοκρατικών θεσμών κτλ. Δηλαδή ε, ε, ε, μια δυσφορία από πλευράς του τύπου σε σχέση με το καθεστώς του Αλκίεφ. Για δε τις αρχές Απριλίου και τα γεγονότα του Τάλλας που εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από πλευράς Ρωσίας τις μέρες εκείνες για μια 100% φορολόγηση του, βαρέ, του πετρελαίου κινήσεως ε, που εξαγόταν προς το Κυργιστάν. Ξαφνικά λοιπόν ανακοινώθηκε ότι επιβάλλεται αυτό ο 100% και βέβαια σε μια χώρα που δεν έχει και στου φυσικού πόρου σήμαινε τεράστια ο οικονομικό ε, άχθο. σήμαινε άμεσο διπλασιασμό κάθε, ε, του κόστους κάθε δραστηριότητας οικονομική και άρα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Τι μπορούμε να πούμε τώρα για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ναι, το όντα απαρτίζεται επιτοπλίστων από πρώην υπουργού, πρώην υπουργού οι οποίοι όμως ε, γρήγορα είδαν, ε, γνώρισαν την απογοήτευση από το καθεστώ του Αλκίεφ και που αρκετά γρήγορα απεμπλάξαν από αυτό. Μάλιστα, ορισμένοι όχι μόνο συμβλήθησαν αλλά και φυλακίστηκαν από το καθεστώ του ΑΛΚΙΕΦ στη συνέχεια. Και άρα, ναι, έχουμε διατηρήσει τι επαφέ μαζί του και ε, το, του στηρίξαμε τα τελευταία πέντε χρόνια με τι παρεμβάσει μα φέτος και τώρα έχοντας ε, εκπροσωπήσει την δημοκρατική αντιπολίτευση στον Αλκίεφ ξέρουν και αναγνωρίζουν πρώτοι αυτοί από κάθε άλλον την παράδοξη θέση, το οξύμορο το οποίο εκπροσωπούν, δηλαδή να είναι και επικριτέ του καθεστώτο και πρώην μέλη του καθεστώτο. Και τώρα αυτό που θέλουν είναι να δημιουργήσουν μια δημοκρατία που να ε, ακολουθεί και τις ιδιαιτερότητες της ε, κυργισικές τρόπον την έτσι ώστε να, έχει ένα προεδρικό, ώστε να ξεφύγουν από το προεδρικό σύστημα των κεντροασιατικών δημοκρατικών με ένα σχέδιο ε, κοινοβουλευτική σταγματική δημοκρατία, δηλαδή με ένα σύνταγμα κοινοβουλευτικό, με πρόεδρο όχι βέβαια μόνο επίτιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει με τι ελάχιστε ε, αρμοδιότητε του προεδρευομένου συστήματο, που θα διαφυλάσει δηλαδή την ακαιρεότητα και την επιβίωση του έθνου, αλλά που πάντως, όπου πάντω ε, την διακυβέρνηση θα την έχει ο Πρωθυπουργό με την κυβέρνησή του, όπω συμβαίνει στα προεδρευόμενα ευρωπαϊκά συστήματα. Αυτό είναι δηλαδή το σύστημα το οποίο διεκδικούν αυτοί οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Μας λένε ότι έχουν την εμπειρία, έχουν αποθαρρυνθεί από το σοσιαλιστικό του παρελθόν και θέλουν να προχωρήσουν πιο σωστά κοινοβουλευτική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτό μας λένε. Πώς ανταποκρίνεται η Ευρώπη. Και εδώ θα προχωρήσω πολύ γρήγορα γιατί δεν χρειάζεται παρά να σας υπενθυμίσω τις βασικές αρχές. Ότι δηλαδή θα θυμάστε ασφαλώς η Λέδη Άστον στις 7, 8 και 9 Απριλίου και μάλιστα στη συγκεκριμένη αυτή ε, περίοδο εγώ είχα αποσταλεί στην Κυργυσία για να απευθύνω και πάλι το μήνυμα που απέστελε η Λέδη Άστον, δηλαδή επάνωδο στην ομαλή ζωή, στην ειρήνη, ε, στην λειτουργία των θεσμών σε μια συνταγματική δημοκρατία, σε ένα συνταγματικό δημοκρατικό καθεστώ και εξού και βρέθηκα παρόν και αυτό τις μάρτυρας των γεγονότων στις 14 και 15 του μήνα στο Μπίσκεκ ε, με μια πολύ καλή προσπάθεια συντονισμού σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη που ξεκίνησε πολύ γρήγορα και νομίζω ότι μπορέσαμε να απευθύνουμε απευθεία το ίδιο μήνυμα στο οποίο αναφέρθηκα και εγώ τώρα μόλις και να επιφτύχουμε μια κάποια επάνωδο στην πολιτική ομαλότητα και τον ορθολογισμό τον πολιτικό και μια ύφεση ίσως ε, σε πρώτη φάση τουλάχιστον με την αποχώρηση του Μπακίεφ, του πρώην Πρόεδρου έτσι ώστε να γυρίσουμε στην ε, ειρήνη, στην εσωτερική ειρήνη. Και ζητούμε συγκεκριμένα μηνύματα φιλοπορίας, για, δηλαδή στάδια επενόδου στην δημοκρατία, όπως ζήτησε και το Υπουργείο των Εξωτερικών, δηλαδή το κείμενο που έχετε λάβει, έχει διανεμηθεί. Και αύριο, ακριβώς το ίδιο μήνυμα, με το ίδιο νόημα, λέει, θα αποστείλουμε στον ε, αναπληρωτή υπουργό, μάλλον στον υπηρεσιακό υπουργό σε μια συνεδρίαση στις Βρυξέλλες με τις Δημοκρατίες Κεντρικής Ασίας για να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις και να το πούμε και εμείς τα μήνυματά μας. Αυτά, Πρόεδρε, σταματώ εδώ και αν μου επιτρέψετε θα μιλήσω μετά στα θέματα της Κεντρικής Ασίας. Αλλά θα προτιμήσω να ακούσω πρώτα τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Δόκτωρα Μορέλ. Κρατήσετε το χρόνο σας. Δεν μακρηγορήσατε. Ε, μοιράζεται ενώ περιμένω δηλαδή να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαρτολότσι, πρόεδρο της αντιπροσωπείας με την Κεντρική Ασία, μοιράζεται έλεγα το πρακτικό για την, ε, το σχετικό πρακτικό μου για την ε, συνάντηση των Υπουργών εχθές. Οπότε θα έχετε επιπλέον πληροφορίες. Πρόεδρε Μπαρτολότσι, έχεις το λόγο. Στα 10 λεπτά όμως, ε. Ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο Αλμπερτίνη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μορέλ, ο οποίος ε, μας περιέγραψε ποια είναι η κατάσταση στην Κυργυζία. Εγώ ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας με την Κεντρική Ασία θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα αυτή την περιοχή λόγω της κατάστασης αλλά και του ενδιαφέροντος, του ρόλου που παίζει αυτή η περιοχή για τη διεθνή ασφάλεια και λόγω των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε αυτή την περιοχή σχετικά με την ενεργειακή προμήθεια. Εγώ παρακολούθησα τα πρόσφατα επεισόδια στην ε, Κυρκυζία και εξέφρασα και τα συλληπιτήριά μου για τα θύματα, εκφράζοντας και την ευχή για την αποφυγή της ε, βίας. Εμείς πριν από πέντε χρόνια θεωρήσαμε ότι η επανάσταση των λοιπόν, δημιούργησε πολλές ελπίδες ε, για το μέλλον ε, της χώρας και θα μπορούσε να επηρεάσει και τις υπόλοιπε χώρες της Κεντρικής Ασίας για να οικοδομήσουν δημοκρατικές κοινωνίες και να παρέχουν καλύτερο βιωτικό επίπεδο και εργασιακό επίπεδο στους πολίτες τους. Οι αρχικές ελπίδες αποδείχθηκαν φρούδες η δυσαρέσκεια του κόσμου αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, οι κατηγορίες ε, για νεποτισμό εκ μέρους ε, της ε, κυβέρνησης και άλλα προβλήματα οδήγησαν στις ταραχές που γνωρίσαμε τις τελευταίες μέρες. Παίζονται όμως στρατηγικά πράγματα σήμερα. Εγώ Είμαι, πέρα από πρόεδρος δηλαδή της αντιπροσωπείας με την Κεντρική Ασία, είμαι και στην, Επιτροπή, στην αντιπροσωπεία, αντιπρόεδρος της με την Κυργυζία. Εμείς ε, πέρυσι είχαμε εκφράσει μεγαλύτερο, ε, το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτής της χώρας. Εμείς θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτεύχθη και γιατί δεν προσεγγίστηκε το απαραίτητο οικονομικό επίπεδο, γιατί υπήρχαν προβλήματα στις μεταφορές και άλλα προβλήματα υποδομών. Πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την αναπτυξιακή βοήθεια. Η στρατηγική για την Κεντρική Ασία πρέπει να λάβει υπόψη όλες αυτές τις πλευρές που αφορούν και στις άλλες χώρες όπως το Τατζικιστάν, το Ουσμπεκιστάν και άλλες και που είναι θεμελιώδης ε, για τη σταθερότητα αυτής της ε, περιοχής της Κεντρικής Ασίας. Για να επιτευχθεί οποιαδήποτε οικονομική ε, επενδυτική δραστηριότητα χρειάζεται σταθερότητα. Χρειάζεται αποκατάσταση του της συνταγματικής νομιμότητας, εκλογές, ελευθεροτυπία, οργάνωση πολιτικών κομμάτων και κοινωνίας των πολιτών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να ε, δράσει ορίζοντας τις απαραίτητες γραμμές σύμφωνα με τις διαδικασίες μας. Και από το ψήφισμα που θα πρέπει να εγκρίνουμε στην επόμενη Ολομέλεια θα πρέπει να τονίσουμε τη βούληση του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να μπορέσουμε συγκεκριμένα να παρέμβουμε σε αυτή την περιοχή που χρειάζεται μια εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να τη βοηθήσει στη σταθεροποίηση μιας πραγματικής δημοκρατίας. Όχι μόνο λοιπόν ευχολογίες αλλά συγκεκριμένες δράσεις. Εγώ όλα αυτά που είδα μέχρι τώρα μου φαίνονται πολύ γενικόλογα, γεμάτα καλές προθέσεις, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Πριν από μερικές ώρες εγώ συνάντησα τον ε, κύριο Αζίροφ, τον πρέσβη της ε, Κυργιζίας και σύμφωνα με τον ε, πρέσβη η προσωρινή κυβέρνηση ελέγχει το σύνολο της χώρας. Και σύμφωνα όμως με τον πρέσβη είναι καμιά τριακοσαριά ε, οπλισμένοι οπαδοί του πρώην ε, Προέδρου με τον οποίο γίνονται διαπραγματεύσεις για να λυθεί η κατάσταση. Η προσωρινή κυβέρνηση, όπως ε, μας είπε και ο, κύριος Μορέλ, πρόβλεψε ένα σχέδιο δράσης για την επάνωδο στη δημοκρατία θα, ε, όπου έχει προβλέψει εκλογές τον Οκτώβριο και το ε, καθεστώς της χώρας θα, γινόταν, θα, θα, θα, θα γίνει πιο κοινοβουλευτικό και λιγότερο προεδρικό. Αυτά αποφάσισε η προσωρινή κυβέρνηση με τους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ. Η επισητιστική προμήθεια στη χώρα είναι σε βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Χρειάζεται να χορηγηθεί επισητιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να παρέμβει η Κομισιόν με ανθρωπιστική βοήθεια για να βοηθήσει τον λαό της Κυργιζίας. Κατά τη γνώμη μου, εγώ δηλαδή υπογράμμισα στον πρέσβη την ευχή να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα ασφαλείας χωρίς να χυθεί περισσότερο αίμα. Και προοδευτική επάνωδο στο δημοκρατικό καθεστώς. Υπογράμμισα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, ε, απέναντι στην, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στην κατάσταση και υποστηρίζει το λαό της Κυργιζίας σε αυτή τη δύσκολη και ιδιαίτερη στιγμή. Αυτή νομίζω ότι πρέπει να είναι και η γραμμή των πολιτικών ομάδων ε, όταν θα καθορίσουν το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει όχι με γενικολογίες αλλά συγκεκριμένα σε μια τόσο σημαντική στιγμή ε, για το λαό της ε, Κυργυζίας ο οποίος ε, αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες. Ευχαριστώ πρόεδρε Μπαρτολότσι. Έχουμε πολλές τοποθετήσεις. Ο κύριος η κυρία Νικολάη, η οποία είναι εισηγήτρια για το Τουρκμενιστάν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αδιαμφισβήτητα έχουμε μία κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική για όλους όσους δηλαδή ενδιαφέρει αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Έχω μπροστά μου τα, συμφέρον, τα συμπεράσματα συγγνώμη, του Συμβουλίου. Και κυρίως η τελευταία παράγραφος Μου φαίνεται λίγο περίεργη, λέει ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση από κοντά στην περιοχή μαζί με τους διεθν ετέρους εταίρους και πρωταγωνιστές. Με αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Πέρα από το ψήφισμα που θα βγάλουμε εμείς, νομίζουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για το πώς θα προχωρήσει στον εκδημοκρατισμό της, στη βοήθεια για τον εκδημοκρατισμό της χώρας για να σταματήσει η βία. Και θέλω να ρωτήσω κάτι το συγκεκριμένο στον κύριο Μορέλ. Λοιπόν, δύο είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές στην περιοχή. Η Ρωσία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτή η προσωρινή κυβέρνηση φαίνεται να έχει ένα πιο συγκεκριμένο δημοκρατικό όραμα. Αλλά όμως και αυτή η προσωρινή κυβέρνηση είναι κομμάτι της παλιάς διοίκησης, του παλιού κατεστημένου. Και υπογράφτηκε φέτος το καλοκαίρι μια συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει αυτές τις χώρες να διαμορφώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα αμερικανικού τύπου ή πιστεύετε ότι αυτές οι χώρες θα πέσουν στα χέρια της Μόσχας. Ευχαριστώ κυρία Νικολάη. Πέτερλε, εισηγητής για το Τζικιστάν. Και ο Ευχαριστώ τον κύριο Μορέλ για την παρουσίασή του. για την κατάσταση στην Κυργυζία. Πριν από πέντε χρόνια παρακολουθούσα από κοντά τα, όσα διαμοιβόντουσαν στην Κυργυζία ως ειδικό απεσταλμένος της Όξε. Και δυστυχώς τα ίδια πράγματα επαναλαμβάνονται. Βέβαια τότε δεν υπήρξε τόση βία, ενώ αυτή τη φορά είχαμε νεκρούς. Η κατάσταση χειροτέρευσε. Δεν υπήρξε καμία δημοκρατική πρόοδος στο μεταξύ. Πόσο μάλλον πρόοδος του κράτους δικαίου. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση δημοκρατικού τύπου σε αυτή τη χώρα. Και τελικά η αντιπολίτευση από πού βγήκε από την προηγούμενη εξουσία, από τους προηγούμενους που είχαν την εξουσία. Ο Μπακύρ είχε συνεργασίτη με τον Αλκάιεφ και ο πρώην υπουργό Εξωτερικών τώρα πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Δηλαδή η ίδια η ΚΙΠ που κυβερνούσε πριν <coughs> παίρνει την κατάσταση στα χέρια της τώρα. Πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση στη χώρα με ιδιαίτερη σοβαρότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει συγκεκριμένα αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνει κανείς την ιστορία αλλά ότι μπορεί κανείς να πράξει ένα ποιοτικό άλμα ένα άλμα προς τα Εμπρό, ένα σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα που σίγουρα θα αλλάξει κάπως τα πράγματα. Αλλά τι θα γίνει μετά, γιατί αυτό ήδη το είχαμε στο παρελθόν αλλά δεν δόθηκε μετά καμία συνέχεια. Σε αυτή τη φάση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί σε μία διαδικασία η οποία δεν θα έχει μόνο ως στόχο τη δημιουργία ενός δημοκρατικού κράτους, αλλά και τις βάσεις εκείνες της διακυβέρνησης αυτού του δημοκρατικού κράτους. Αυτή η χώρα, ακόμη και αν είναι μικρή, είναι πάρα πολύ σημαντική για τη σταθερότητα. Δεν είναι σημαντικό το αν έχει πετρέλαιο ή δεν έχει πετρέλαιο. Εγώ πιστεύω ότι η στρατηγική μας για την Κεντρική Ασία πρέπει να έχει μια εξέχουσα θέση. Πριν από πέντε χρόνια δεν είχαμε έναν ειδικό αντιπρόσωπο σε αυτή τη χώρα, τώρα τον έχουμε. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια περιοχή για την οποία χρειάζεται να προσέχουμε ιδιαίτερα για να αποφύγουμε τα προβλήματα στο μέλλον. Προβέρα, πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ρωτήσω τον πρέσβη Μορέλ που τον ευχαριστώ για την έκθεση. Υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε υποψίες α, ε, ε, θρησκευτικής ε, θρησκευτικών εξτρεμιστών στην περιοχή και Ισλαμικής παρέμβασης εσείς επίσης πιστεύετε ότι με ένα νέο σύνταγμα μπορούμε να ορίσουμε ε, ε, ένα κοινοβουλευτικό καθεστώς. Πιστεύετε ότι αυτές οι θεσμικές αλλαγές μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση αν δεν εργαστούμε επί της ε, κοινωνικής και συλλογικής συνείδησης ούτως ώστε ο κόσμος να αλλάξει ο λαός να αλλάξει, δηλαδή μήπως πρέπει να γίνει μια προσπάθεια δηλαδή και στην κοινωνία των πολιτών και στην παιδεία για να έχουμε μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα, πράγματα δηλαδή που είναι πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ κύριε Προβέρα. Βαϊντέρε, κυρία Βαϊντέρε. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, καθώς επίσης και με τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Άστον. Θεωρώ ότι οι δηλώσει αυτέ ήταν ιδιαίτερα γενικόλογε, χρησιμοποιούσαν κάποιε συνηθισμένε εκφράσει. Λέγαμε ότι θέλαμε να εξασφαλίσουμε τη δημοκρατία. Πολύ καλέ οι προθέσει αυτέ. Δυστυχώ όμω δεν μα λένε τίποτα το ουσιώδε. Θα ήθελα να είχα απαντήσει σε κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει που μεταλανίζουν. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η στάση που έχουμε απέναντι στην προσωρινή κυβέρνηση. και ποια είναι η στάση της μεταβατική αυτής κυβέρνησης σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, το προηγούμενο καθεστώς. Ο κύριο Μωράτη μα είπε ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση στη Ρωσία αναφέρθηκαν πάρα πολύ έντονα στι εξεγέρσει ε, στη Κυργυζία και το ίδιο έγινε και για την Γεωργία, δηλαδή αντιτάχθηκαν πάρα πολλά μέσα μαζική ενημέρωση εναντίον τη ε, Γεωργία. Μου προκαλούν ανησυχία τα γενικότερα σχόλια τα οποία έγιναν εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντίδραση στα σχόλια αυτά. Βλέπουμε ότι στα πλαίσια της εξέγερσης αυτής στην Κυργυζία υπάρχουν ε, πολλοί διαδηλωτές που έχουν ε, κλέψει όπλα και οπλοφορούν αυτή τη στιγμή. Και είναι ανησυχητικό αυτή τη στιγμή ότι διαπραγματεύσεις γίνονται με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για το πρόεδρο στο παρελθόν. Ποια θα είναι λοιπόν η στάση μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αποδεχθούμε την προσωρινή αυτή κυβέρνηση, την μεταβατική αυτή κυβέρνηση. Και πώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με μια στεναρή φωνή. Αν απλώς ακολουθούμε τα γεγονότα άβουλα, θεωρώ ότι δεν θα καταφέρουμε να επέμβουμε σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική από στρατηγική πλευρά. Ευχαριστώ. Mm, eh, Ευχαριστώ κυρία Βαϊντέρη. Η κυρία Νεβεγκάλοβα. Ευχαριστώ πολύ. Μου δίνετε το λόγο. Πρώτη ερώτηση ή μάλλον καταρχάς να εκφράσω τι ευχαριστίε μου στον κύριο Μορέλ για την έκθεσή του. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι γνώστη των πραγμάτων. Έχει ασχοληθεί εντατικά με το θέμα αυτό και θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια περιοχή με πολλούς παράγοντες, με πολλές συνισταμένες θα πρέπει να, λάβουμε, να εξετάσουμε ιδιαίτερη σοβαρότητα και προσοχή. Ερωτώ λοιπόν τι θέλει να, τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και προς για να βελτιώσει την κατάσταση. Δεν θέλω μόνο ωραία λόγια παρακαλώ, ότι χρειάζεται να βοηθήσουμε κτλ. Συγκεκριμένα μέτρα. Τι έχετε υπόψη. Υπάρχει δυνατότητα παραδείγματι να διατεθούν κονδύλια, υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης ανθρωπιστικού ανθρωπιστικής βοήθειας ή κάποιων δραστηριοτήτων ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για περιοχή που ε, είναι ασταθής, το λιγότερο, συνορεύει με το Αφγανιστάν, πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε δράση ουσιαστική. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να διακόψουμε ίσως τις ε, τοποθετήσεις να μιλήσετε εσείς για να συνεχίσουν με τα υπόλοιποι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές για τις εύστοχες ερωτήσεις τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με μεγάλη σαφήνεια, μόνο ότι θα προσπαθήσω να είμαι και σύντομος για να ακούσουμε και άλλους ε, ομιλητές, να συνεχιστεί η ανταλλαγή απόψεων δηλαδή. Όσον αφορά την παρέμβαση του κυρίου ε, Μπαρτολότσι που αναφέρθηκε στο κέντρο διέλευσης, στο σταθμό διέλευσης του Μανάς. Σίγουρα το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σαφώς αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα σταθμό διέλευσης όλων των συστημάτων των στρατιωτικών, είτε πρόκειται για εξοπλισμούς, είτε πρόκειται για προσωπικό, ε, και έχει να κάνει ουσιαστικά με την παρουσία του Αμερικανικού στρατού στο Αφγανιστάν ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια ζώνη κοντά στο αεροδρόμιο του Μπισκέκ. Η ζώνη αυτή ονομάζεται Μανά. Στο παρελθόν ήταν στρατιωτική βάση και μετά τις συμφωνίες του Ιουνίου ονομάζεται πλέον σταθμός διέλευσης. 500 με 600 άτομα κάθε μέρα προσγειώνονται στο σταθμό αυτό και ετοιμάζονται να πάνε στο Αφγανιστάν ή επιστρέφουν μετά το τέλος της αποστολής τους από το Αφγανιστάν και κάνουν ένα διάλειμμα, μια παύση στο σταθμό αυτό προτού γυρίσουν στις χώρες τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για μια βάση πάρα πολύ στρατηγική για όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις, για όλους ουσιαστικά τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπλέκονται στρατιωτικά στο Αφγανιστάν. Μας αφορά λοιπόν άμεσα, μεσότατα η βάση αυτή και είμαστε ακόμα πιο σαφείς. το στρατηγικό δίκτυο των ΗΠΑ θα τους επέτρεπε να έχουν και άλλους διάβλους πρόσβαση στο Αφγανιστάν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο εύκολα αν δεν υπήρχε αυτός ο σταθμός ανεφοδιασμού, αυτός ο σταθμός διέλευσης. Πήγα δύο φορές στην βάση αυτή και μπορώ να σας πω ότι πραγματικά μπορούμε να δούμε μόνο και μόνο από την όψη τους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν στο Αφγανιστάν και αυτούς οι οποίοι επιστρέφουν από το Αφγανιστάν. Τους τελευταίους μήνες η Ισπανία και η Γαλλία στείλανε δυνάμεις στρατοτικές αλλά και ιατρικές προς το Αφγανιστάν και έγινε επίσης στη βάση αυτή ένας πολύ σημαντικός ανεφοδιασμός όσον αφορά τις γαλλικές στρατοτικές δυνάμεις. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες νεφοδιασμού και στις γειτονικέ περιοχές. Παρ' όλα αυτά η βάση Μανάς παραμένει πάρα πολύ σημαντική και είναι η πιο κεντρική βάση. Κυρία Νικολάη στη συνέχεια. Κίνα, Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία σίγουρα είναι βασική εταίρεια. Μην ξεχνάμε όμω και την Κίνα, την οποία ανέφερα. Η Κίνα βρίσκεται πολύ κοντά στην Κυργυζία. Είναι πολύ σημαντικό παράγοντα λοιπόν στην ε, ισορροπία τη ε, χώρα αυτή και συμβάλλει και από οικονομική ε, πλευρά γιατί ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η Κυργυζία αποτελεί τον ε, τόπο διέλευσης των κινέζικων εξαγωγών προς την Κεντρική Ασία. Και αυτό για να ολοκληρώσουμε λοιπόν την εικόνα των όμορων χωρών. Τώρα, αμερικανικό μοντέλο και ρωσικό μοντέλο. Δεν θα ήθελα να σας απαντήσω ευρωπαϊκό μοντέλο στην ερώτησή σας, πάντως πρέπει να σας πω ότι ε, η επιλογή που γίνεται αυτή τη στιγμή από τους ηθήνοντες είναι μια κοινοβουλευτική επιλογή. Το βλέπουμε αυτό ήδη σε επιλογές που κάνουν στις εργασίες τους. Ουσιαστικά χρειάζονται τη βοήθεια της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης προκειμένου να καταφέρουν να περάσουν προς μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Θα γίνει μια εργασία μέχρι τις 18 ε, Μαΐου και ε, στη συνέχεια θα ξαναπάω επιτόπου μέσω της ανανεωμένης εντολής που μου έχει δοθεί από την Κάθριν Άστον και συμφωνήσαμε χθε με τον ε, γραμματέα της Επιτροπής της Βενετίας η Επιτροπή της Βενετίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης να έχουν κοινή στάση. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί την παρέμβαση της Επιτροπής της Βενετίας επιτόπου και ο κύριος Μαρκέρτ, το Γενικός Γραμματέας Επιτροπής Βενετίας που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα των Βαλκανίων, θα ξεκινήσει τις ε, εργασίες υποστήριξης που θα γίνουν από το Συμβούλιο της Ευρώπης από τις 6 Μαΐου και μετά θα αποσταλούν από τις 11 Μαΐου και μετά εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα συμμετέχουν και αυτοί στις εργασίες που θα γίνουν επί τόπου και θα έχουν ως στόχο να παρέχουν, να παρέχουν συμβουλές και να υποστηρίξουν την δημοκρατική διαδικασία στη χώρα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη δική μας πολιτική εμπειρογνωμοσύνη μετά από το αίτημα του Κυργιστάν, το αίτημα βοηθείας προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινοβουλευτική δημοκρατία στη χώρα αυτή. Τώρα σε σχέση με τις άλλες ερωτήσεις ε, που θέσατε. Η Κυργισία αποτελεί μια χώρα που βοηθά πάρα πολύ την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στον Βόρειο και τον Νότιο Κάυκασο. Θέλουμε να βοηθήσουμε το σύνολο λοιπόν της χώρας και όχι μόνο συγκεκριμένε περιοχές της χώρας αυτής. Προκειμένου να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος, θα πρέπει να καταφέρουμε να τονώσουμε την εθνική διάσταση της χώρας. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να περάσουμε στη δημιουργία εθνικών πολιτικών κομμάτων και να έχουμε πραγματικούς καταλόγους ε, εκλογικούς προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την εθνική αυτή διάσταση. Τα τελευταία 20 χρόνια μέσω της ε, προεδρευόμενης δημοκρατίας στην Κυργυζία είδαμε τελικά ότι η ύπαρξη ενός μόνου βασικού αυταρχικού κόμματος έχει δημιουργήσει συνθήκες νεποτισμού που δεν βοηθούσαν καθόλου την δημοκρατική διαδικασία στη χώρα. Προκειμένου λοιπόν να εκφραστεί σωστά δημοκρατικά από πολιτική πλευράς η χώρα χρειάζεται τη δική μας υποστήριξη, υποστήριξη τόσο πολιτική όσο και οικονομική και θα πρέπει να καταφέρουμε από το σύνολο της Ευρώπης, από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωση, να στείλουμε τους καλύτερους εμπειρογνώμονέ μας. Στη συνέχεια, όσον αφορά τα μέλη της προσωρινής εκείνης κυβέρνησης οι οποίοι συμμετείχαν στην προηγούμενη κυβέρνηση, στο προηγούμενο καθεστώς. Ναι, όντως, αλλά πρόκειται για άτομα τα οποία πέρασαν πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή ακριβώς επειδή επέλεξαν να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον πρόεδρο Μπακίγεφ. Σίγουρα αυτό θα αποτελεί απόλυτη εγγύηση για το μέλλον. Σαφώς θα πρέπει να στείλουμε τα σωστά μηνύματα επιτόπου, τα οποία είπατε και εσείς. Αυτό όμως προσπαθούμε να κάνουμε και σας διαβεβαίω, αυτό κάνουμε σε καθημερινή βάση και τονίζουμε κάθε φορά τις προσδοκίες τις οποίες έχουμε από την Κυργυζία. Αύριο, για παράδειγμα, ένας από τους υπηρεσιακούς υπουργού θα πρέπει να μας δώσει τις απαραίτητες διασφαλίσεις όσον αφορά την ελευθεροτυπία, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού στις ε, φυλακές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εργαζόμαστε πλέον για πάρα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και πετούμε πλέον αποτελέσματα για τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα και διασφαλίσεις. Τώρα, όσον αφορά την νέα γενιά και τα άτομα τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες κυβερνήσεις, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί απέναντί τους. Υπάρχει, αν θέλετε, η τρίτη αυτή δύναμη που ουσιαστικά είναι άτομα τα οποία εργάζονται για πολιτιστικούς συλλόγους, για αθλητικούς συλλόγους, που ουσιαστικά όμως ε, προωθούν άλλες πεπιθήσεις ε, και ουσιαστικά κάνουν εντελώ διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία διατείνονται ότι κάνουν και σίγουρα οι πεπιθήσεις τους δεν είναι απαραίτητα πάντα δημοκρατικές. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί απέναντι στα νέα αυτά πρόσωπα. Τώρα, ο κίνδυνος του φονταμενταλισμού σαφώς υπάρχει. Έχουμε όμως και μία κοινωνία των πολιτών πλέον στην Κυργυζία. Έχουμε ένα οικογενειακό κοινωνιολογικό Ισλάμ και όχι θεολογικό Ισλάμ στη χώρα αυτή. Εξισλαμίστηκε η Κυργυζία σχετικά αργά. Ήταν ε, ένας νομαδικός λαός αρχικά. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την, το Ισλάμ στην Κυργυζία με τον τρόπο που εκφράζεται το Ισλάμ σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Η Κυργύζη είναι ένας νομαδικός βουνίσιος λαός που δημιουργήθηκε και εγκαταστάθηκε στην περιοχή αυτή τον 19ο αιώνα. Πρόκειται λοιπόν για ανθρώπους με έντονες απεπιθήσεις, αν θέλετε, στην ε, οικογένεια, σε κάποιες αξίες καθημερινής ζωής και δεν ακολουθούν ε, με δογματισμό τις αρχές του Ισλαμισμού. Θεωρώ ότι ακόμα και η ε, θρησκεία στη χώρα αυτή εξασκείται με τρόπο καθαρά ειρηνικό. Τα τελευταία όμω χρόνια έχουμε δει ότι όντω υπάρχουν εξτρεμιστέ οι οποίοι ασκούν πίεση στην χώρα αυτή. Διάφορα κινήματα, κινήματα ταμπλήρ και άλλα που έρχονται από εξωτερικές χώρες έχουν προσπαθήσει να ρίζοσπαστικοποιήσουν το Ισλάμ στην Κυργιζία. Ως πρεσβευτής το 1992 επισκέφθηκα πολλές από τις ζώνες της Κυργιζίας και πρόσφατα έλαβα την ε, επιβεβαίωση ότι ε, όντως έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι, α, τάσεις αυτές από εξωτερικές χώρες της α, Κυργιζίας. ουσιαστικά η άνοδος αυτή του Ισλαμισμού έχει να κάνει με τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού, με τις πολύ δύσκολες καθημερινές συνθήκες που πρέπει να αντιμετωπίσουν ε, οι πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι η Κυργυζία είναι μια χώρα με πολύ αντίξωες συνθήκες, με ένα πολύ κρύο κλίμα. Ε, είναι πολύ εύκολο λοιπόν δυσαρεστημένοι πολίτες να πέσουν στην παγίδα του ε, εξτρεμισμού. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι στις ε, εξελίξεις αυτές. Κάποιες άλλες ερωτήσεις τώρα που μου θέσατε. Ποια είναι η στάση μας, αν είναι επαρκή σε αυτή τη στιγμή η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο χθε έδωσε έναν προσανατολισμό, επιβεβαίωσε την αρχική μας δέσμευση, ήμασταν από την αρχή παρόντες επιτόπου, στείλαμε συγκεκριμένα και ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα από την αρχή. Είπαμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε μια ειρηνική έξοδο από την κρίση αυτή. Θελήσαμε να καταφέρουμε να εδραιώσουμε μια πάρα πολύ ασταθή ειρήνη και αύριο θα επιβεβαιώσουμε τα μηνύματα αυτά και θα, θα αρχίσουμε μάλλον την συνεργασία μας με τους ε, υπουργούς της ε, προσωρινής μεταβατικής αυτής κυβέρνησης της ε, Κυργιζίας. Τώρα όσον αφορά την χρηματοδότηση και αυτό το ζήτημα μας απασχολεί. Απαντώ στην κυρία Νεβίντοβα, 30 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή μπορούμε να δώσουμε. Το πιο σημαντικό είναι τα χρήματα αυτά βέβαια να φτάσουν επί τόπου. Παρά την κρίση που πλήττει τη χώρα, θα πρέπει τα χρήματα αυτά να φτάσουν επί τόπου. Εδώ και πάνω από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί 300.000 Κυργιζίους οι οποίοι ζουν στην πιο μειονεκτούσα περιοχή της ε, χώρας, στην νότια δηλαδή Κυργιζία, στην κοιλάδα του Φεργανά. Σαφώς θα πρέπει να συνεχιστεί η υποστήριξη αυτή χρηματοδοτική από ανθρωπιστική τώρα πλευράς. Δεν υπάρχουν κάποιες επίγουσες ανάγκες, ότι πήγαμε στην Κυργυζία την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε ότι θα πρέπει να ερευνήσουμε περισσότερο ποιες είναι οι άμεσες ανάγκες και ποιες θα πρέπει να είναι οι άμεσες δράσεις μας που θα οδηγήσουν στην σταθεροποίηση της ε, χώρας. Ελπίζω να πάνε σε ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ, δόκτωρα Μορέλ. Έχουμε προβλήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμά μας για σήμερα. Πρέπει να ολοκληρώνω τις τοποθετήσεις με τους τέσσερις εγγεγραμμένους. Τελευταίο τμήμα λοιπόν, τελευταίος γύρος συζητήσεων. Η κυρία Γέγκελ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Μουρέλ. Δεν θα τα χρειαστώ τα τρία λεπτά. Μας ε, δείξατε κύριε Μουρέλ ότι έχετε βαθύτερη γνώση της περιοχής και ιδιαίτερα τη Κυριακή. Και ότι μεριμνείτε ιδιαίτερα για την περιοχή αυτή. Ερωτώ λοιπόν, πολύ συγκεκριμένα, μπορείτε να απαντήσετε. Αρκούν τα μέσα που έχουμε στη θέση μα. Αρκούν τα μέσα ώστε το όντι να ανατραπεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση. Όταν ε, εξελέγει πριν από πέντε χρόνια ο Μπακίεφ, θεωρήσαμε ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Και για αρκετό διάστημα παρακολουθούσαμε να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο δυστυχώ. Υπήρχαν τα μηνύματα δηλαδή αρκετά νωρί. Τώρα, με επισητιστική βοήθεια ή με χρήματα που ενδεχομένω θα μπορούσαμε να προσφέρουμε αν και θα σα υπενθυμίσω ότι και πριν από δύο ή τρία χρόνια είχαμε διαθέσει ακόμα 300.000 ευρώ σε πιστιστικη βοήθεια, 300 εκατομμύρια ευρώ σε επιστηστική βοήθεια. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί θα πρέπει να παραλάβουμε κάτι το οποίο είδαμε ότι δεν βοήθησε τον πληθυσμό στην ουσία, τον λαό στην ουσία. Τι θα κάνουμε τώρα, τι διαφορετικό και καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Ε, πολιτική, εκδημοκρατισμό, ανθρωπιστική βοήθεια, ναι, είναι πολύ σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό από όλα νομίζω είναι να συμβάλλουμε ώστε να ε, εξασφαλιστεί η συμβίωση, η ειρηνική συμβίωση του Βορρά με τον πολύ φτωχότερο νότο της χώρας. Τη χώρα τη γνωρίζω εγώ αρκετά καλά, την παρακολουθώ 10-10 χρόνια. Βλέπω όμως ότι δεν έχουμε κινηθεί εγκαίρως στα ουσιαστικά ζητήματα και γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο σε σχέση με τις ε, ε, ασιατικές δημοκρατίες, κεντροασιατικέ δημοκρατίες αναλάβει μια δραστηριότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση με, την, με σταθερή παρουσία, ίσως με μόνιμο ε, γραφείο εκεί πέρα. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσω για το Ισλάμ το οποίο αναφέρατε νωρίτερα ως παράγοντα της πολιτικής ζωή, Ναι, αλλά και τη συμφωνώ μέσα θεωρώ ότι η φτώχεια που επικρατεί στον Νότο μπορεί να αποτελέσει πηγή για άλλες εξελίξεις και να επηρεάσει διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γέγκελ. Κύριος Μπόρης. Και εγώ ε, είμαι μέλος της Επιτροπής ε, της Αντιπροσωπείας για την Κεντρική Ασία. Μα αυτό το οποίο είδαμε είναι τελικά συνδεδεμένο με την αδυναμία του κράτους και της οικονομίας. Το είδαμε και στο παρελθόν, το βλέπουμε και τώρα. Θέλω όμως να κάνω μια γενική παρατήρηση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πολιτική της για την Κεντρική Ασία. Η Κυργυζία δεν θα πρέπει να αποτελεί απόδειξη της ουσιαστικής στράτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική Ασία για να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο λαμβάνοντας επίσης ότι ανταγωνιστές μας στην περιοχή είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία έχουμε 20 χρόνια εμπειρίας για, την τη δημοκρατική οικοδόμηση και θεωρούμε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην βοήθεια που δίνουμε για τον εκδημοκρατισμό και στην ε, βοήθεια που δίνουμε για στην ολοκλήρωση των ε, μεταρρυθμίσεων. Αυτή η στρατηγική θα είναι σοβαρή και συνεχής ή θα είναι πρόσκαιρη. Κύριος Δόρφμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πολύ γρήγορες ερωτήσεις στον κύριο, σύντομες συγγνώμη ερωτήσεις στον κύριο Μορέλ. Πώς εκτιμάτε τη σταθερότητα της χώρας σε αυτήν τη φάση Υπάρχει κίνδυνος επαναφοράς της βίας, ε, στη βία και πώς αξιολογείτε εσείς ε, την κατάσταση εν ώψη αυτού του συνταγματικού δημοψηφίσματος η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα πάλι της βίας ε, ή πιστεύετε ότι είναι κάτι που όλος ο κόσμος συμμερίζεται η Κομισιόν αν θέλει το λόγο, μπορεί να μιλήσει για τρία λεπτά και αν δεν θέλει το λόγο να δώσουμε το λόγο στον δόκτορα Μορέλ για τα συμπεράσματα. Πολύ, Πολύ σύντομα πρόεδρε. Μια και εκπροσωπώ την ε, Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας στην ΕΚΟ και δεν μπορώ να κάνω σχόλια για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια θα μιλήσω. Όπως γνωρίζετε δεν είναι σύστημα διαχείρισης πολιτικών κρίσεων, ο κύριος Μορέρα, δεν το διατύπωσε ξεκάθαρα. Υπάρχει εκπρόσωπος μας στον Μπισκέικ ε, Πιτόπου δηλαδή, ο οποίος αναλύει την κατάσταση, έχει υποβάλει και μια πρώτη έκθεση που δημοσιεύτηκε, μάλλον ε, διανεμήθηκε στα θεσμικά όργανα και στα κράτη-μέλη, σήμερα το πρωί μάλιστα και η οποία έκθεση λέει ουσιαστικά ότι οι κύριες ανθρωπιστικές ανάγκες, οι οποίες είναι λιγότερο οξυμένες αυτή τη στιγμή, έχουν καλυφθεί. Και ότι οι εταίροι με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ συχνά είναι σε θέση να ανταποκριθούν και με ίδιους πόρους στις ανάγκες που προκύπτουν από την ανθρωπιστική κρίση. Αλλά πάντα είμαστε, στη θέση, δηλαδή είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αν χρειαστεί αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Ολοκληρώνει ο Δόκτωρ Μορέλ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια ερώτηση στην οποία δεν απάντησα και είναι σημαντική. Αναγνωρίζουμε ή όχι τη νέα αυτή κυβέρνηση. Πολύ συχνά μας κάνουν την ερώτηση αυτή, ασχοληθήκαμε με αυτήν από την αρχή. Η οχι την που κάναμε είναι ξεκάθαρη από την αρχή δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα αναγνώριση κυβέρνηση αυτή. Αναγνώριση αυτή καθ' αυτή. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Από το να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή με τι νομικέ διαστάσει μια προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση, αυτό το οποίο θα πρέπει να σα απασχολήσει περισσότερο είναι η σταθεροποίηση τη χώρα αρκεί βέβαια η κατεύθυνση που ακολουθείται αυτή τη στιγμή να είναι η σωστή. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στείλαμε από την πρώτη στιγμή. Και αυτό επιβεβαίωσε και η Κάθριν Άστον, μολονότι ορισμένοι μπορεί να θεωρούν ότι οι δηλώσεις, δηλώσεις της ήταν γενικόλογες. Πάντως το μήνυμα ακούστηκε με απόλυτη σαφήνεια στην BISCEC και περιμένουμε αύριο συγκεκριμένε απαντήσεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα να κινηθούμε με τον τρόπο αυτό από το να ασχολούμαστε κυρίως με τυπικότητες στη στιγμή που η κατάσταση είναι πάρα πολύ ασταθής και ευάλωτη. Πρέπει να γίνει τους επόμενους έξι μήνες μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Το είπε και αυτό και το είπαν και προαλήσαντες. Έχουμε το δημοψήφισμα τον Ιούνιο και τις εκλογές στη συνέχεια τον Οκτώβριο. Τώρα, Ακούστηκαν κάποιες ερωτήσεις για τις ε, επιτόπου ανάγκες και για το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί. Η εμπειρία καταδεικνύει και το είπε αυτό και ο εκπρόσωπος της ε, ΕΚΟ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εγκαθιδρύσουμε το κράτος δικαίου, ακόμα και να αυτό σημαίνει να οικοδομήσουμε νέες φυλακές, γιατί το σφρονιστικό σύστημα βρισκόταν πραγματικά σε μια άθλια κατάσταση. Θέλουμε επίσης να τροποποιήσουμε το ποινικό κώδικα και να επιφέρουμε όλες τις απαραίτητες αυτές αλλαγές προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν τόπου οι βασικοί προσανατολισμοί που επιλέξαμε από την αρχή. Και ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σταθερότητα στη χώρα είναι η απασχόληση των νέων, καθώς επίσης και η δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας. Επιγόντως λοιπόν χρειάζονται προγράμματα κυρίως γύρω από τον Μπισκέκ. Πρέπει να καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε την περιοχή γύρω από το Μπισκέκ, μια περιοχή που πλήττεται από ανεργία της τάξης του 30-40%, τόσο πολύ βέβαια πολλές φορές απαντάτε στις ορεινές περιοχές όπως το Ναρίν. Καταλαβαίνετε όμως ότι η υψηλή αυτή ανεργία οδηγεί σε δυσαρέσκεια, σε αγανάκτηση και πάρα πολλοί νέοι στρέφονται σιγά σιγά προς την προς το έγκλημα, προς τα δίκτυα παράνομης ε, εμπορίας και διακίνησης. Και κάτι ακόμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε για την Κυργυζία είναι ότι υπάρχει μια πολύ καλά διαρθρωμένη παράνομη παράπλευρη οικονομία. Μια μαύρη οικονομία. Και καταλαβαίνετε ότι ε, γίνονται αυτή τη στιγμή και νέες απόπειρες προκειμένου να εγκαθιδρυθεί εκ νέου ένα νέο εγκληματικό δίκτυο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εργαστούμε με τις ε, αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να καταφέρουμε να πατάξουμε την εγκληματικότητα και τη διακίνηση των ε, ναρκωτικών. ελοχεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι και ουσιαστικά πάρα πολύ στα πλαίσια της αστάθειας αυτής που χαρακτηρίζει τη χώρα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες που ενδεχομένω να τους δοθούν για να προχωρήσουν σε νέες παράνομες δραστηριότητες. Αναφέρθηκα πριν από λίγο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει επί τόπου και στην πρώτη μου έκθεση, μετά την πρώτη μου επίσκεψη στο Μπισκέκ, είχα πει ότι ε, θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να έρθουν στην Ευρώπη, ιδίως στους νέους αυτούς που ζουν σε αντίξωες συνθήκες, που δεν έχουν δουλειά, που έχουν αγανακτισμένοι. Προβλέπεται συνεργασία με τα πανεπιστήμια, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Erasmus Mundus. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται επί τόπου Απαντώ έτσι στον στην κυρία Ζιγγέλ. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται επιτόπου η πρέσβης κυρία Στεμπέλ βρίσκεται επιτόπου και, έχουμε, και έχει γύρω της μία, ένα πλήρες επιτελείο. Με τη βοήθεια του Συμβουλίου αποστήλαμε εμπειρογνώμονες προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες πολιτικές αναλύσεις από μια ομάδα που βρίσκεται επί τόπου. Βλέπετε λοιπόν ότι η Επιτροπή είναι επί τόπου. Πρέπει απλώς να ενταθεί η εργασία αυτή τη στιγμή. Η ε, Γερμανία που έχει μια πλήρως λειτουργούσα πρεσβεία εκπροσωπεί ουσιαστικά και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργό Εξωτερικών τη Γαλλία ε, Κουσνέρ μα είπε επίση ότι και η Γαλλία θα ανοίξει μία πλήρως λειτουργούσα πρεσβεία στο Μπισκέκ. Το παράδοξο είναι ότι ε, η χώρα αυτή που βρίσκεται τόσο κοντά τελικά στην Ευρώπη είναι μια πλήρω οποία δεν εκπροσωπείται η Ευρώπη. Νομίζω ότι και αυτό το παραδοξο ειναι οτι η χωρα αυτη που βρισκεται τοσο κοντα τελικα στην ευρωπη ειναι μια χωρα στην οποια δεν εκπροσωπεί το η ευρωπη νομιζω οτι και αυτο το μηνυμα θα πρέπει να το στείλουμε προ όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αναλάβουν τι ευθύνε του. Τώρα, όσον αφορά το νότιο τμήμα τη χώρα. Όντω τίθεται το ζήτημα αυτό δεν θα πρέπει όμως να επιμένουμε πάρα πολύ. Φοβηθήκαμε κάποια στιγμή ότι θα διαχωριστεί η χώρα. Ο Νότος με τον κύριο Μπακίγεφ θα υποστήριζε τον κύριο Μπακίγεφ και ότι ο Βοράς θα υποστήριζε την προσωρινή κυβέρνηση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ο ίδιος ο Νότος της χώρας, ο πληθυσμός εκεί, είναι απογοητευμένος από τον κύριο Μπακίγεφ. Στο Τζαλαλαμπάντ, για παράδειγμα, που βρίσκεται στον, στη Νότιο Κυργιζία, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι. Ο Στάλιν μάλιστα είχε διαχωρίσει την κοιλάδα που βρίσκεται στην νότιο περιοχή της χώρας, δίνοντας το ένα στο Σβεγγιστάν, το άλλο κομμάτι στο Τατζικιστάν. Ήταν μια τεχνική διαίρεση, αν θέλετε, και βλέπουμε ακόμα μια τεχνική διέρη και βασίλευε και βλέπουμε ακόμα και τις συνέπειες σήμερα. Ενδεχομένω ο κύριος Μπακίγεφ να περίμενε θα έχει την υποστήριξη του Νότου. Δεν συμβαίνει όμω κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα ακολουθήσει οτιδήποτε κάνει το Μπισκέκ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η προσωρινή κυβέρνηση να μείνει σε επαφή με όλες τις δυνάμεις της χώρας και να μην μπει σε ένα παιχνίδι εσωτερικής πολιτικής. είναι πολύ σημαντικό η μεταβατική κυβέρνηση να είναι σε θέση να αφουγκραστεί το σύνολο των δυνάμεων παντού στη χώρα. Και μέσω της εκπόνησης του νέου συντάγματος ακριβώς αυτό επιθυμούν να επιτύχουν, να καταφέρουν ουσιαστικά να εκπροσωπήσουν το σύνολο των δυνάμεων της χώρας. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ε, όλοι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν θέλουν να προκαταλάβουν τις καταστάσεις. Είδαμε πάντως με τις διαδηλώσεις τελευταίων ημερών ότι ε, η κατάσταση μπορεί να πάσα στιγμή να κλιμακωθεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα καθεστώς, μια κατάσταση εθνικής ενότητας, προκειμένου η κατάσταση να μην ε, κλιμακωθεί Στην, στα προάστια του Μπισκέκ είχαμε θανάτους πέντε ατόμων και κατευθείαν υπόθηκε ότι επρόκειτο για άτομα κουρδικής καταγωγής. Προσπάθησαν σαστικά να δώσουν μια πολιτική διάσταση στην, στα γεγονότα αυτά. Ουσιαστικά επρόκειτο για μικρές ομάδες ανθρώπων από μειονότητες που είχαν εγκατασταθεί έξω από το ΒΙΣΚΕΚ και ουσιαστικά ήταν μια μικρή εγκληματική ομάδα, ουσιαστικά ήταν μαφιόζοι και προσπάθησαν κατευθείαν να χαρακτηρίσουν τις μικρές αυτές ομάδες εγκληματών ως εθνοτικές ομάδες, ως μειονότητες. Σαφώς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτική και ο εκπρόσωπος του ΑΣΕ, ο απεσταλμένος του ΑΣΕ βρίσκεται στην ε, Μπισκέκ και εργάζεται στα πλαίσια του Πνεύματος Επιτροπής της Βενετίας και θέλει να δει πώς θα εκπροσωπηθούν στο νέο κοινοβουλευτικό σύστημα οι μειονότητες. Αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουμε και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δίνουμε υπερβολικές διαστάσεις σε ένα πρόβλημα το οποίο μέχρι στιγμής ήταν ε, ελεγχόμενο. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες ε, βίες διαδηλώσεις, η κατάσταση όμως παραμένει ευάλωτη. Για παράδειγμα, για το δημοψήφισμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα κρίση θα πρέπει να γίνει με απόλυτη διαφάνεια θα πρέπει να, γίνεται υπό την, να γίνει υπό την επιτήρηση της διεθνούς κοινότητας προκειμένου η όλη διαδικασία της ψηφοφορίας να εξελιχθεί α, ομαλά. Αυτό ισχύει τόσο για το δημοψήφισμα όσο και για τις εκλογές που θα ακολουθήσουν. Σαφώς στο παρελθόν και το γνωρίζουμε αυτό από τις αποστολές του ΟΑΣΕ ότι υπήρχε πολύ σημαντικό περιθώριο βελτίωσης. Θα ολοκληρώσω λίγο την παρέμβασή μου όσον αφορά την Κεντρική Ασία, την ευρύτερη περιοχή. Προσπαθούμε να επανεξετάσουμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2007 για την Κεντρική Ασία Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η στρατηγική μας εκεί. συμμετέχουν ομάδες από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξ αρχής είχαμε δεσμευτεί ότι πρόκειται να θεωρήσουμε τη στρατηγική αυτή. Δεν πρόκειται να αλλάξει εντελώς η στάση μας και να ακολουθήσουμε εντελώς διαφορετικό δρόμο. Πρέπει απλώς να είμαστε επικριτικοί, να αξιολογήσουμε την στρατηγική αυτή και να πούμε ουσιαστικά ότι εμπλουτίστηκε η στρατηγική αυτή τα τελευταία χρόνια το τελευταίο διάστημα έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ την διάσταση της ασφάλειας στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής, προσπαθώντας να καλύψουμε εξελίξεις σε χώρες όπως το Ιράν. Προσπαθούμε να έχουμε ένα πιο έντονο διάλογο όσον αφορά τα θέματα της ασφάλειας. Το ζήτημα του ύδατος επίσης, του νερού, πήρε πάρα πολύ σημαντική διάσταση στα πλαίσια της στρατηγικής μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προωθήσει μια περιφερειακή συνεργασία για το νερό. Επίσης, η διαχείριση των συνόρων. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, γιατί μόνο αυτό θα καταφέρει να συμβάλλει στην απόλυτη ασφάλεια των χωρών αυτών και αυτό θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Επανεξετάζουμε λοιπόν τη στρατηγική μας, θέλουμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η Κυργυζία μας δίνει τώρα τη δυνατότητα να καταφέρουμε να αξιολογήσουμε πιο αυστηρά μετά από τρία χρόνια την στρατηγική μας. Η δυναμική υπάρχει όμως. Σε πάρα πολλούς τομείς καταφέραμε να πάμε πιο μακριά περιμένουμε, από ό,τι περιμέναμε. Μην ξεχνάτε ότι ήταν μετά την επανάσταση της ε, Τουλίπας που αποφάσισε η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει έναν ειδικό εντεταλμένο στην ε, περιοχή. Το Μάρτιο του 2005 ήταν τα γεγονότα στο Μπισκέκ που μας κάνανε να εντατικοποιήσουμε και να ξεκινήσουμε τη στρατηγική στην περιοχή αυτή. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε βέβαια στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, έχουμε την υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να δημιουργήσουμε πέντε αντιπροσωπείες επιτόπου, δηλαδή επιπλέον στον Τατζικιστάν, το Ουσβεκιστάν και το Τουρκμενιστάν, χώρες στις οποίες δεν υπάρχει ακόμα εκπροσώπηση. Ο πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει τελικά για την δημιουργία της εκπροσώπησης αυτής. Αυτό που μας ενδιαφέρει να καταφέρουμε να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα στο σύνολο των χωρών της περιοχής. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι μερικά από τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο. Και θα έλεγα τέλο ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την πολιτική διάσταση των σχέσεών μα. Οι περιοχέ αυτέ ε, είναι ρωσόφωνες κυρίω. Αυτό ε, δικαιολογείται απόλυτα από ιστορική ε, πλευρά. Δεν θα πρέπει όμω η επικοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι μόνο από τη Ρωσία. Και ένα πάρα πολύ θετικό παράδειγμα είναι ότι επιτόπου ο πληθυσμός μπορεί πλέον να παρακολουθεί τις ειδήσει του Euronews. Ε, μόνο και μόνο αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Το κόσμο μπορεί και να ενημερώνεται μέσα από το Euronews. Αυτά είχα να σα πω. Έτσι θα ακολουθήσουμε τη στρατηγική μα τα περισσότερα χρόνια. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ακριβέστατη απάντησή σας, Δόκτωρα Μορέλ. Ευχαριστώ πολύ είχαμε τις απαραίτητες πληροφορίες και μπορέσαμε να έχουμε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα και πλήρης. Λοιπόν, θα μείνετε μαζί μας και για το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και αυτό με την ιδιότητά σας ως εκπρόσωπος, ειδικός εκπρόσωπος της Ένωσης για την κρίση στη Γεωργία. Παρακαλώ. Μάλλον ευχαριστώ τον πρόεδρο Μπαρτολότσι για την παρουσίασή του και καλό τον δόκτωρα Σέμπι να έρθει στο βήμα να μας μιλήσει για το επόμενο θέμα. Έχουμε λοιπόν την έκθεση της Κομισιόν για την... είναι η έκθεση από την επίσκεψη της Αντιπροσωπείας Επιτροπής ε, Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας στην Τυφλίδα. Θα ακούσουμε λοιπόν την έκθεση του Προέδρου. Συνάντησαν εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφους ε, και γενικά ε, ε, κατάφεραν και πήγανε στα σύνορα με την Οσετία. Δίνω το λόγο στον κύριο Τάλερ και μετά οι ειδικοί εκπρόσωποι μπορούν να μιλήσουν οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν. Μετά βέβαια από την πρώτη τοποθέτηση. Αν περιοριστείτε στα 8, maximum 10 λεπτά, θα μου επιτρέψετε να κλείσω τα επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης εγκαίρως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και επιτρέψτε μου να είμαι σύντομος αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο επίπεδα της έκθεσης. Θα αναφερθώ δηλαδή πρώτα στο, στα τεθέντα και δεύτερον σε διδάγματα που θα πρέπει να αντλήσουμε από την επίσκεψη στην Τυφλίδα. Έγινε δηλαδή η 12η συνεδρίαση της Αντιπροσωπής Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας στις 29 με 31 Μαρτίου στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Τέσσερις ευρωβουλευτές, όχι πολλοί δηλαδή, μόνο τέσσερις. Αλλά το πρόγραμμα ημερήσια διάταξη, οι επισκέψεις ήταν όλα πολύ εντατικά. Οι συζητήσεις με τους γεωργιανούς ομολόγους μας επικεντρώθηκαν καταρχάς στο λεγόμενο δεύτερο κύμα δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, τις επερχόμενες δημοκρατικές εκλογές που όπως γνωρίζετε θα έλαβαν χώρα στις... Θα λάβουν χώρα στις 30 Μαΐου, τοπικές εκλογές. Ε, μετά έχουμε να συζητήσουμε, είχαμε να συζητήσουμε την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τον τρόπο με τον οποίο οι Γεωργιανοί αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτής. Θέματα εθνωτικών μειονοτήτων, εσωτερικός εκτοπισθέντων και προσφύγων. και επιπλέον ε, το, τα διοικητικά σύνορα και τη διαχείριση αυτών με την Νότια και την προοπτική των συνομιλίων στη Γενέβη. Επίσης, με εταιρική σχέση συζητήθηκε, συζητήσαμε την Περιφερειακή ε, συνεργασία στην ε, περιοχή του Εύξηνου Πόντου και του Νότιου Κάφκασου, καταλήξαμε σε ε, δηλώσεις και συστάσεις, πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει το Δεκέμβριο με την αντιπροσωπεία του Αζερβαϊτζάν, θα θυμάστε ίσως κάποιοι εξημών. Και θα θυμάστε ίσως. Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ξεκινήσαμε και μια μεγάλη συνεδρίαση με παρουσία πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπροσώπων του τύπου, εκπροσώπων τη αντιπολίτευση, που μα ενημέρωσαν για την προετοιμασία και τα διάφορα ζητήματα που ε, έχουν, είναι επικαιρότητα, ζητήματα ώψη των τοπικών εκλογών ε, εξέφρασαν οι κυβερνητικέ οργανώσει και οι υπόλοιποι παριστάμενοι επικρίσει και ως προς την κατάσταση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πλουραλισμού, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δυνατότητα να συμμετέχουν ε, κατά τρόπο ισότιμο και δίκαιο στις τοπικές εκλογές. Καταλήξαμε σε κοινό συμπέρασμα ότι η απρόσκοπτη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών σε συνδυασμό με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου αποτελούν κρίσιμη σημασία ε, όρους για την ε, λειτουργία της ε, γεωργίας, για την γεωργία στη σύγχρονη εποχή. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να συναντηθούμε και με τον πρόεδρο Σακασβίλη, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, καθώς και άλλους αξιωματούχους της γεωργίας. Είχαμε επίσης και την ευκαιρία, τελευταία ημέρα της αποστολή μας εκεί, να συναντηθούμε, να επισκεφθούμε μάλλον την Ευρωπαϊκή Μονάδα Παρακολούθησης ε, της κατάστασης στη Γεωργία. Ακούσαμε τις απόψεις τους και για τα διοικητικά σύνορα που ξέρετε ότι μετά τον Αύγουστο του 2008 και τον πόλεμο με τη Ρωσία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Επισκεφθήκαμε τον Κόρνη συναντηθήκα με τους ιστορικούς, εκτοπιστέντες και πρόσφυγες, τον Τίτη Κουρβαλέτη, ένα στρατόπεδο προσφύγων που βρίσκεται πολύ κοντά ε, με τα διοικητικά σύνορα της ε, περιοχής του Συρβάλη. Πιο σημαντικό όμως, και θα ήθελα εδώ ακριβώς να συγκεντρωθώ, είναι να δούμε τα διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από τις συζητήσεις μας και σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούμε πάντα στη Γεωργία. Καταρχάς λοιπόν, η κατάσταση στα διοικητικά σύνορα της Νότιας Ουσιατίας και της Απχαζίας είναι ήρεμη εδώ και μερικούς μήνες. Ιδιαίτερες εξελίξεις στις συνομιλίες της Γενέβης μεταξύ των εμπλεκομένων στη σύρεξη ε, πλευρών δεν υπάρχουν. Εξελίξεις από πλευράς της ε, ε, αποστολής παρακολούθησης, εποπτείας μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει. Δεν επιτρέπεται όμως αυτή την αποστολή να περνάει από την άλλη μεριά εκεί που ελέγχουν ε, τα εδάφη οι Ρώσοι. Δηλαδή μόνο από την πλευρά της Γεωργίας μπορεί να κοιτάξει την κατάσταση αυτή η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν οι πρώτες ε, Δημοκρατικέ εκλογέ, μάλλον γίνονται οι πρώτε δημοκρατικέ εκλογέ, 30 Μαου, με χαρακτήρα ιδιαίτερα σημαντικό γιατί δεν είναι κοινέ τοπικέ εκλογέ. Έχουμε να κάνουμε μέχρι και με την εκλογή δημάρχου για, το, για την Τυφλίδα. Ε, αλλά πάνω από όλα η σημασία του είναι ότι μέχρι το 2012 που έχουμε τι πρώτες γενικές εκλογές και το 2013 που προβλέπονται οι προεδρικές εκλογέ, δεν, δεν υπάρχουν άλλε, Δηλαδή είναι τοπικέ εκλογέ σήμερα και θα ξαναγίνουν σε δύο χρόνια πάλι εκλογέ. Και έτσι η κατάσταση είναι αυτή, είναι τέτοια που φαίνεται πως ορισμένα μέσα και ορισμένες πολιτικές δυνάμεις προσπαθούν να ασκήσουν πίεση με την χρήση των κάποιων εξωτερικών δυνάμεων στο εσωτερικό. Θα ακούσατε ίσως για μια εκπομπή πρόσφατα ένα ε, ντοκιμαντέρ, ε, ψευδεπίγραφο όμως, 30 λεπτό, για μια λεγόμενη νέα εισβολή την οποία είχε υποστηρίξει η αντιπολίτευση της Γεωργίας. Και εκεί όταν ήμασταν επί τόπου ενημερωθήκαμε ότι ο κόσμος πανικοβλήθηκε όταν έμαθε τέτοια πράγματα, όταν είδε τον ντοκιμαντέρ αυτών, Υπήρχαν και αποβολές ακόμη εγγύων γυναικών και ε, καρδιακές προσβολές. Και βέβαια κατεβλήθηκε η προσπάθεια να, και από δική μας πλευράς να ηρεμήσει η κατάσταση. Τέτοιες πιέσεις λοιπόν και εντάσεις, οι οποίες ασφαλώς ε, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από, το, αυτό που επιδιώκει η δική μας ε, αποστολή παρακολούθησης και πτήρησης κατάστασης, δηλαδή την εξομάλυνση των συνθήκων και την ειρήνευση. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία της Γεωργίας δεν θέλουν να προξενούν φόβους ε, και να εκφοβίζουν ή ε, να κατατρομοκρατούν το λαό, αλλά θέλουν να προχωρήσουν προς μια ομαλή κοινοβουλευτική δημοκρατία κτλ. Υπάρχει βέβαια περιθώριο για ανάπτυξη ρωσικού τύπου για ανάπτυξη μάλλον περισσότερων ε, διαφορετικών πολιτικών κομμάτων και όχι μόνο ρωσικού τύπου πολιτικής εξουσίας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί να βοηθήσει και ο τύπος. Επιπλέον, ζωτική σημασία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ιδιαίτερη παρουσία και κύρος στη Γεωργία, να ασκήσει αυτό κύρος. Η Γεωργία είναι ένας από τους μεγαλύτερους, ε, από τα κράτη που έχουν περισσότερο ωφέλεια, στηρίζονται ιδιαίτερα στην οικονομική μας βοήθεια και την παρουσία μας εκεί. Αυτό άλλωστε καταγράφεται και στην κοινή μας δήλωση με τους Ιωριανούς. Εν τέλει δεν σημειώνω ότι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Γεωργία έχει μεγάλη σημασία και ιδιαίτερα την, ε, για την διατήρηση, για την προστασία μάλλον και επίτευξη των στόχων και της ασφάλειας ε, στις ε, προμήθειες ενέργεια τη γεωργία πρέπει να τη δούμε ως χώρα συνολικά και όχι μόνο ως αρχές, επίσημες αρχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στόχος και θα πρέπει να τον επιδιώξουμε από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τάλερ. Ο κύριος Τσαρνέκη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολούθησα την ε, τοποθέτηση του συναδέρφου Τάλερ. Πιστεύω όπως και στην Σλοβενία η τηλεόραση, το ραδιόφωνο μπορεί να παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον ε, πρόγραμμα και ανάλογα αν αρέσει ή δεν αρέσει ο κόσμος το κοιτάει. Στη Γεωργία τι έγινε τελικά παρουσιάστηκε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σε μια τηλεόραση που δεν ήταν κυβερνητική τηλεόραση και έγινε όλη αυτή η φασαρία. Σκεφτείτε όμως εσείς τι έγινε και στη Νέα Υόρκη. Τότε η στη δεκαετία του 30 η εκπομπή του Orson Welles ε, όπου προσωμείωθηκε ε, μια επίθεση αριανών. Τι θα γινότανε τότε, ποιον θα καταδίκασαν την κυβέρνηση ή το ραδιοφωνικό σταθμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι οι σταθμοί τελικά κάνουν πολλά πράγματα για να αυξήσουν την ακροματικότητα. Δεν πρέπει εμείς λοιπόν να κριτικάρουμε τον πρόεδρο Σακασβίλη για αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ πάντως με τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας και λέω ότι πρέπει να διατηρήσουμε ουσιαστική βοήθεια για τη Γεωργία που σίγουρα ε, δικαιούται αυτή τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι είναι μια χώρα η οποία στέκεται δίπλα μας αποφάσισε καθαρά και εξάστερα να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίθετα με την Αρμενία βγήκε από την οικονομικό πολιτική επιρροή της Ρωσίας και γι' αυτό και τιμωρήθηκε. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα. Και η χώρα έχει μία κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ εγώ κύριε Μορέλ για την ε, ειλικρίνειά σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα στην Κυργυζία. είναι δυναμική, είπαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε μια γερμανική πρεσβεία, θα ανοίξει και μια γαλλική πρεσβεία. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση πιο συνολικά. Ο κύριος Χατζή Γεωργίου, για δύο λεπτά. ότι εμείς και νομίζω ότι όλον το σώμα πρέπει να υποστηρίξουμε την ανεξαρτησία και την ακαιρεότητα της γεωργίας θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να είναι θεμελιώδες για τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στις εξελίξεις εκεί και βεβαίω πρέπει να υποστηρίξουμε ότι πρέπει κανείς να αποφύγει οποιασδήποτε στρατιωτικές ενέργειες προς την α ή την β κατεύθυνση και να δούμε αν μπορεί και πώς μπορεί να επιληθεί το ζήτημα με ειρηνικά μέσα. Έχω δύο ερωτήσεις. Ε, πώς κρίνεται ότι θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών, το α αποτέλεσμα ή το β αποτέλεσμα της πολιτικής εξελίξης, όχι τον εκδημοκρατισμό της χώρας, αλλά τις οποιασδήποτε πολιτικές εξελίξεις και κάτι συναφές στην Απχαζία και την Οσετία θα υπάρχουν εκλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χατζηγεωργίου. Η κυρία Λέζινγκ για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ. Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ε, έκθεση Επιτροπής Κοινοβουλευτική συνεργασία. διάβασα και την έκθεση. Αναφέρεστε στην έκθεση αυτή στη δημιουργία μιας νέας διεθνούς ε, ομάδας ε, επιβολής της διατήρηση διατήρησης ειρήνη. Πότε θα δοθεί όμως πλήρης εντολή στη αυτή δύναμη και θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι η γνώμη της Ρωσίας για την πρόταση αυτή. Στην έκθεση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας επικρίνεται σε κάποια σημεία πολύ σφοδρά η Ρωσία. Σε κάνα σημείο την επικρίνεται η Γεωργία. Μολονότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι η Γεωργία είναι αυτή που ξεκίνησε τον πόλεμο. Θεωρείται λοιπόν ότι μεροληπτεί κάπως η έκθεση. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά σε κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας στην έκθεση, μολονότι η αμερικανική πλευρά παρέχει και κατάρτιση στις α, γεωργιανές στρατιωτικές δυνάμεις. Για ποιο λόγο δεν γίνεται, γίνεται σχετική μνήμα στην έκθεση. και για ποιο λόγο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε σχέση με, την, με το αίτημα της Αμερικανικής Γερουσίας να συνεργαστεί μαζί της και η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξοπλιστούν εκ νέου οι ε, γεωργιανοί στρατιώτες. Και επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιους παραλληλισμούς ανάμεσα στη Γεωργία και το Κωσυφοπαίδιο. Ευχαριστώ κύριο Λέζινγκ. Κλείνουν οι τοποθετήσει. Αφήνω το λόγο στον δόκτωρα Μορέλ. Διότι μου είπαν ότι πρέπει σύντομα να φύγει. Δηλαδή στις 5 θα φύγει. Και θα θέλαμε να μάθουμε πέρα από τις απαντήσεις και ορισμένες πληροφορίες στα πλαίσια του διαλόγου της Γενέβης κυρίως ε, ενώ, ε, στα όσα μισολάβησαν συνεδρίες στις 30 Α, κύριε Λούνατσεκ, θέλετε το λόγο? Ένα λεπτό, κύριε Λούνατσεκ, όμως. Α, κυρία Λούνατσεκ, συγγνώμη, επειδή είστε εισηγήτρια. Α, δεν είστε εισηγήτρια. Ήσασταν όμως παρούσα στην αντιπροσωπεία. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Όχι, δεν είμαι συγγήτρια για τη Γεωργία. Ήμουν όμως μέρος της αντιπροσωπείας, της επίσκεψης που α, κάναμε με την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας. Δεν ήμουν στο πρώτο τμήμα της συζήτησης, δεν ξέρω πόσα πράγματα έχετε καλύψει. Το πιο σημαντικό πράγμα που είδαμε κατά την επίσκεψή μας είναι ότι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική ότι θα πρέπει να τη βελτιώσουμε, να την ενισχύσουμε, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πληθυσμούς και στις περιοχές της Νοτιού Οσετίας. Ένα άλλο σημείο το οποίο εμεί είδαμε αρκετά ως αρκετά προβληματικό είναι η διαδικασία με την οποία πρόκειται να γίνουν οι εκλογές, το ότι άλεξαν κάπως οι εκλογικές περιφέρειες, ιδίως γύρω από την Τυφλίδα. Επίσης, ε, τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένα κόμματα όπως το Πράσινο Κόμμα στην ε, χώρα, μας είπαν ότι δεν μπορούσαν να καταχωρηθούν στους καταλόγους τους εκλογικούς, δεν μπορούσαν να καταγραφούν για τις ε, εκλογές και ότι ήταν ε, μάλλον ότι οι εφορευτικές ε, επιτροπές ε, αποτελόντουσαν από κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εκπροσώπους της κυβέρνησης. Πράγμα το οποίο καθιστά, όπως καταλαβαίνετε, τις εκλογές ιδιαίτερα μεροληπτικές, όχι ανεξάρτητες και αυτό το πρόβλημα το είχαν τονίσει και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επίσης, στην εκπόνηση των εφορευτικών επιτροπών, στην σύστασή τους, ορισμένοι εκπρόσωποι από μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν είχαν γίνει δεκτοί. Επίσης, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης είχαν επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν, είχαν επικρίνει την... Είχαν αναφερθεί στο πόσο δύσκολο ουσιαστικά είναι να καταφέρουν να εκπέμπουν κάποιοι σταθμοί και το ζήτημα αυτό το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Σακασβίλη, ο οποίος μας είπε ότι ναι, γνώριζε ότι ε, υπήρχαν επικρίσεις για τα ζητήματα αυτά. Είναι σημαντικό λοιπόν, πέρα από οτιδήποτε κάνουμε, να υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος βαθμός ε, αυτοκριτικής στη χώρα αυτή. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα, καταφέρει, θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα με το Κοινοβούλιο της Γεωργίας, νομίζω το γνωρίζετε αυτό. Πιστεύω πάντως ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταφέρουμε να, παρακολουθήσουμε εκ του σύνογγες εξελίξεις στη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λούνετσεκ. Ο κύριος Μορέλ, 5-6 λεπτά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήδη μίλησα πολύ. Θα είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνεται να απαντήσω σε αυτά που υπόθηκαν για την αποστολή ε, την οποία παρακολούθησα με ενδιαφέρον. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε μία δράση ε, και να πω όσα αρμόζουν στη δική μου, στο δικό μου ρόλο, σε, αυτή, δηλαδή, σε αυτές τις συζητήσεις της ε, Γενέβης. Εμείς συνεργαζόμαστε με τον συνάδελφο, βρισκόμαστε στον ίδιο όροφο στη Ρίντε Λαλουά, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες μας με αποστολή την συζητήσεις ε, της ε, Γενέβης και λυπούμε που δεν μπόρεσα να δω συγκεκριμένες αναφορές στις συζητήσεις της Γενέβης που αποτελούν τμήμα του γεωργιανού ζητήματος. Η αποστολή ήταν επιτόπου ε, και είναι πολύ σύντομη αναφορά στις συζητήσεις ε, της Γενέβης και αυτός είναι ο δρόμος όπου, που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ΟΗΕ ε, για την εξέβρεση μιας διεξόδου μετά από την σύγκρουση σύντομη μένα αλλά πολύ αποσταθεροποιητική Τη δε του 2008. Εμείς ε, στις 30 Μαρτίου που αναφέρατε κύριε Πρόεδρε ήμασταν ε, στο 10ο γύρο συζητήσεων και τα πράγματα ε, προχωράνε και γιατί στην αρχή είχαμε το αίσθημα ότι θα σταματούσε, θα μπλοκαριζόταν η κατάσταση και θα ήμασταν σαν διέξοδο. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζονται οι συζητήσεις, προχωρούμε σταδιακά και αργά μένα, αλλά σταδιακά αργά γιατί βγαίνουμε από έναν πόλεμο ε, όπου η απόρριψη ήταν ολική και από τα δύο μέρη και είμαστε σε μια κατάσταση πολύ πολύπλοκη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την αναγνώριση μιας χώρας ε, που μέγα ποσοστό της παγκόσμιας κοινότητας δεν αναγνωρίζει κλπ. Εμείς ε, θελήσαμε να εξασφαλίσουμε ένα μίνιμουμ βιωτικό επίπεδου στους ε, πληθυσμούς της περιοχής, να ξαναφτιάξουμε ένα καθαστός ασφάλειας και μετά από αυτό να ξεκινήσουμε τις πιο πολιτικές επιλογές. Με υπομονή καταφέραμε με τη μέθοδο του από το, από το ειδικό στο γενικότερο, από το κάτω προς τα πάνω, να ξεκινήσουμε κάτι. Ε, δηλαδή είδαμε εμείς ε, στις λεπτομέρειες ε, τι χρειάζεται ο κόσμος κλπ. Και, και σιγά σιγά ανεβήκαμε επίπεδο. Αυτά για να δημιουργηθεί και ένας μηχανισμός πρόληψης των διαφόρων επεισοδίων. Είτε είχαμε να κάνουμε με την Απκαζία, είτε με την Οσετία, είτε με τη Γεωργία. Πήγαμε καλύτερα με την Απκαζία, με το Τσιμβαλί πήγαμε λιγότερο καλά. Εμείς ως συμπρόεδροι πηγαίνουμε επί τόπου, κοιτάμε να εξετάζουμε την ε, κατάσταση των ε, γεωργιανών ε, μειονοτήτων, επισκεπτόμαστε χωριά προσφύγων, διαπιστώνουμε την κατάσταση επί τόπου, είτε πάμε στο Σουχούμι ή δουλειά λοιπόν που γίνεται στη Γενέβη γίνεται σιγά σιγά, η ομάδα ε, δουλεύει συλλογικά, έχουμε καμιά εξινταριά ε, συμμετέχονται σε όλη αυτή τη διεργασία και βασιζόμαστε στην αποστολή παρακολούθησης Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει δεσμευτεί σε αυτόν τον μηχανισμό πρόληψης των επεισοδίων και προς προσπαθεί να εμποδίσει επεισόδια. Δεν έχουμε την, πλέον την παρουσία του ΟΗΕ και δεν υπάρχει και ο ΑΣΕ. Σιγά σιγά λοιπόν εμείς ε, έχουμε πάρει την κατάσταση στα χέρια μας, είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι στην κατάσταση ε, στην Γεωργία και διασφαλίζουμε και τη γραμματεία στη Γενέβη. Τώρα, έτσι όπως έχει η κατάσταση. Το να παίζει κανείς αυτού του είδους τα σενάρια είναι σαν να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Και η, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε θέση. Έπρεπε να αντιδράσουμε άμεσα και στα 10 λεπτά που επακολούθησαν η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία ήταν αυτή που είπε «Στοπ, δεν τρέχει τίποτα» και ξεφούσκωσε αυτό το γενικό κλίμα ε, πανικού. Πρόβλεψη και ρύθμιση των επεισοδίων. Αυτό είναι απαραίτητο. Εμείς θα πρέπει να ποτίσουμε φορτιμήσεις στους 350 αυτής της αποστολής που αναλαμβάνουν καθημερινούς κινδύνους με τις ε, άλλες 27 χώρες αποστολής. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά τους, αλλά πρέπει πέρα από αυτά να οικοδομήσουμε πριν λάβουμε θέση για την ε, για την ε, για το επεισόδιο το οποίο έγινε μας είπανε ορίστε πρέπει να καταδικάζετε. Ε, εμείς πήραμε θέση και η ΟΑΣΕ και ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαμε όχι. Αν καταφέρνουν, όταν κάτι, ένα επεισόδιο οδηγεί στη δημιουργία ενός πανικού αυτού του μεγέθους, είναι γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται από την άλλη μεριά. Οπότε εμείς στη Γενέβη τι θελήσαμε να παλέψουμε. Να παλέψουμε στη συλλογή των πληροφοριών στην Γενέβη, να μαζεύουμε στοιχεία, Και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει το ρόλο της και είναι πολύ χρήσιμη. Αυτά τα 60 άτομα συνεδριάζουν μηνιαίως και προσπαθούν να δώσουν ένα κλίμα, να δημιουργήσουν ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αυτά για να σας αναφέρω το ρόλο που παίζουν οι συζητήσεις στη Γενέβη. Αυτός είναι λοιπόν ο άξονας ε, γύρω από τον οποίο γυρίζουμε. Τώρα κυρία Λούνατσεκ, εμείς, ε, εγώ ε, διάβασα την ε, τροπολογία σας και για το θέμα της διοικητικής γραμμής διαχωρισμού μιλάει για να σιδηρούν παραπέτασμα. Το καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των ε, πληθυσμών που βία ε, διαχωρίστηκαν. Λοιπόν, ο, ο ποταμός είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως όριο και κόβει, ε, και την κοιλάδα στα δύο. Και Όταν ας πούμε κάποιος έχει επιλέξει να στέλνει τα παιδιά του από την άλλη όχθη του, ε, του ποταμού έχει πρόβλημα να περάσει και έχουμε μία ε, ένα βίο διαχωρισμό χωριά που κόβονται στα δύο κλπ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε λοιπόν εμείς τα περάσματα, να καταπολεμήσουμε την ε, εγκληματικότητα, ε, και να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο δυνατότητες ομαλής διαβίωσης. Και είπαμε θα δημιουργήσουμε εθνικά σύνορα με τη βοήθεια των ε, Ρώσων. και θέλουμε εμείς όταν ορίζονται αυτά τα σύνορα να μπορέσουμε να το κάνουμε με γνώμονα τη διευκόλυνση των πολιτών. ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, πολύ συγκεκριμένες οι απαντήσεις. Εσείς ε, είπατε ότι πρέπει να φύγετε κατά τις 5, σας ε, χαιρετάμε από τώρα, μπορείτε να μείνετε όμως μαζί μας μέχρι σας χάτων και μετά να φύγετε, να στρίψετε αλλά αγγλικά, λέει ο πρόεδρος. Ο πρέσβης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις, καταρχάς. Έχει εξορροπηθεί αρκετά η κατάσταση στο Νότιο Κάφκασο εν γέννη, ειδικότερα στην ε, Γεωργία. Τα διαφιλονικούμενα ζητήματα έχουν και στρατηγικό βέβαια χαρακτήρα και πιο ειδικό. Σε στρατηγικό επίπεδο η κατάσταση είναι η εξής, ότι η Γεωργία έχει να κάνει μια επιλογή και γίνεται βέβαια η συζήτηση της πολιτικής γραμμής που θα ακολουθήσουμε, δηλαδή προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο, για περισσότερη ασφάλεια και ευημερία. Θα πρέπει δηλαδή να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφετέρου δε, ως άλλη επιλογή, αυτή μιας πολιτικής πιο αυτάρκους, μια πιο αυτάρκης γεωργία. διότι ορισμένοι θεωρούν ότι μια ευρωπαϊκή λύση, η φιλοευρωπαϊκή λύση, θα δέσει τα χέρια των ε, κυβερνώντων στη Ρωσία. Ειδικά μέσα σε μια περίοδο που θεωρούν οι κυβερνώντες, οι θύνοντες ε, και η κυβέρνηση ειδικότερα, ότι δεν αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γεωργία. Ένα παράδειγμα ήταν αυτό το ντοκιμαντέρ, του ψευδεπίγραφου ντοκιμαντέρ περί υποτιθέμενου πολέμου. Ένα άλλο θέμα που έχει λίγο πολύ, που πρέπει να κρυθεί λίγο πολύ τώρα, είναι η μοίρα της ε, Δημοκρατίας της Γεωργίας, η οποία τώρα έχει, όπως ξέρετε, ε, στο εγγύς μέλλον τις τοπικές δημοτικές εκλογές, οι οποίες έχουν προσλάβει ασυνήθιστη συμμαχησία. Πρόκειται για μια πρόβα πριν από τις γενικές και προεδρικές εκλογές που προβλέπονται σε δύο-τρία χρόνια. Πρόκειται για εκλογές δημοτικές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ύστερα από την πιο ταραγμένη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας της Γεωργίας με τα προβλήματα του 2007 ε, στην ενέργεια, το 2008 τον πόλεμο, τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια που κράτησαν τρεις μήνες το 2009. Και βεβαίω τίθεται το ερώτημα εάν θα επιτρέπει το γενικότερο πολιτικό κλίμα τη διεξαγωγή ε, ανώθευτων και δίκαιων εκλογών, αλλά και εάν μετά τι εκλογέ θα ε, αποδεχθεί η εξουσία το, ε, την ετοιμιγορία της κάλπης. Και αυτό θα το πρέπει να το δούμε όπως έχουμε αντιμετωπίσει και τις άλλες πολιτικές κρίσεις του 2007 και του 2009. Ένα άλλο θέμα, τρίτο θέμα, οι περιοχές των συγκρούσεων, για τις οποίες έχει γίνει λόγος πολλής, όπου και πάλι θα πρέπει να εξηγήσουμε απλουστευτικά ότι η επιλογή, το δίλημα για την γεωργία είναι ή να απομονώσει αυτές τις περιοχές κατά τρόπον ώστε να ξεχαστούν λίγο πολύ ή να προχωρήσει σε πιο αποφασιστική ε, δράση και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την επίλυση των προβλημάτων και των σειράξεων, που όμως ως λύση δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται στα δικά μας αυτιά. Καθήκον δικό μας είναι να στηρίξουμε τα πιο ε, φωτισμένα μυαλά και στην Τυφλίδα, αλλά και από την άλλη πλευρά των συνόρων. Έχουμε κάνει τις προσπάθειές μας ήδη στο σκοπό αυτό με την Επιτροπή για την Εσωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια που συζήτησε στα τέλη του 2009 μια πολιτική, ένα έγγραφο μάλλον πολιτικής που ε, ε, απαριθμούσε τις διάφορες παραμέτρους για την ε, ειρήνευση και την ασφάλεια στην Οσετία και την Απχασία. με στόχο να ενισχυθούν οι τοπικοί πληθυσμοί κατά τρόπον ώστε να φτάσουν το χειρότερο δυνατό προς την επίλυση των συγκρούσεων, να υπά... να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ιστορικών εκτοπιστέντων και να εξασφαλιστεί συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα πέραν των διοικητικών συνόρων και συμπεδών της Ουσιατίας και Απχαζίας. Και πάλι εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με κενά της εν που πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί ε, το να υπάρξει εμπλοκή χωρίς αναγνώριση της, ε, ε, των θέσεων της άλλης πλευράς μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο επικίνδυνα από τις τελέσματα. Και έχουμε επίσης προχωρήσει σε προσφορά υπηρεσιών, συμβουλών δηλαδή προς την Γεωργιανή κυβέρνηση για το πώς μπορούν να χειριστούν τα θέματα των λεγόμενων κατεχωμένων εδαφών, ένα πρόγραμμα δράσης για το πώς μπορούν να χειριστούν τα ζητήματα αυτά και τώρα υπάρχει μια συμβουλευτική επιτροπή η οποία έχει ε, επιλεγεί ακριβώς για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού και με δεδομένες τις ε, επαφές ε, και με, με την Τυφλίδα και με τις περιοχές των συγκρούσεων όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Τέταρτο σημείο που θα πρέπει να συνυπολογιστεί είναι οι σχέσεις της Γεωργίας με τους γειτονές της. Εκ των φυσικά η μεγαλύτερη χώρα είναι η Ρωσία. Είναι η χώρα που παρουσιάζεται την πιο περίπλοκη εικόνα προς τις σχέσεις με τη Γεωργία, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι βρίσκεται σε στασιμότητα η κατάσταση, διότι δεν εκπληρούνται οι δεσμεύσεις περί καταπαύσης του πυρός. Και υπάρχουν μόνο κάποιες αμυδρές προσπάθειες για βελτίωση των σχέσεων, άνοιγμα δηλαδή ενός μεθοριακού σταθμού μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Στοιχεία όμως ε, μάλλον περιορισμένης απήχησης, κάποιες μικρές επαφές, περιορισμένες επαφές ενώ ταυτόχρονα υπάρχει δυσπιστία και κυρίως από πλευράς της Γεωργίας βλέπουμε τις αντιδράσεις ορισμένων και από την αντιπολίτευση ε, της Γεωργίας. Μάλιστα υπήρξαν φόβοι σε επίπεδο Γεωργίας ότι η Ρωσία μπορεί να ετοιμάζεται για μια νέα επιθετική πολιτική. Σχέσεις με την Τουρκία επίσης έχουν βαρύ ιστορικό. Η Τουρκία είναι στρατηγικός και απαραίτητος εταίρος της Γεωργίας. μένα. Υπάρχουν όμως εντάσεις, ιδιαίτερα λόγω των σχέσεων της Τουρκίας με την Απχασία, την συνεχιζόμενη αποστολή ε, υλικού, εμπορίου δηλαδή, συνεχιζόμενου εμπορίου ε, μεταξύ Τουρκίας και Απχαζίας, με κάποια επεισόδια που έλαβαν χώρα το τελευταίο καλοκαίρι. και τα οποία εξωθούν σε ακρότες μερικές φορές ε, και μέλη της διασποράς της Αυχασίας που είναι αρκετά ισχυρή στην ε, ε, Τουρκία. Έτσι λοιπόν έχουμε την προσπάθεια από πλευράς μας να προωθήσουμε τις συμφωνίες ελευθεροπορίου, ελεύθερων συναλλαγών, συμφωνίας εμπορίου που είναι το καλύτερο μέσον για μας να πιέσουμε προς βελτίωση της κατάστασης και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε, εάν τα πράγματα πάνε καλά, να τις υλοποιήσουμε ως προς τη δημοκρατία. Πρέπει να προσπαθήσουμε, όπως έγινε και, με τις άλλες, και στις άλλες περιπτώσεις του παρελθόν, και να δείξουμε ότι ναι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Παραμένει καυτός ο φάκελος αυτός, η Γεωργία δηλαδή, και ίσως να μην είναι τόσο θετικές εξελίξεις όπως θα τις θέλαμε, αλλά πάντως θα πρέπει να εμείνουμε στο να είναι θετικές και να επιμείνουμε να έχουμε παρουσία και στις αποσχιστήσεις περιοχές και να βοηθήσουμε την άλλη πλευρά να εμπλεκεί στις διαπραγματεύσεις και συνομιλίες και να διαφυλάξουμε την ασφάλεια, μάλιστα στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος παράγων στην περιοχή αυτή, ο κύριος παράγων, ο κύριος παράγων που διαφυλάσσει την ασφάλεια και τις σταθερότητα, είναι η κατάσταση αρκετά δύσκολη. Με την αποστολή της, με την επιστολή παρα, ε, επιτήρησης και τις συνομιλίες της Γενέβης. Δεν θα επεκταθώ. Θα κάλυψε ο κύριος Μορέλ αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ehm, eh, Ευχαριστούμε πολύ τον ε, πρέσβη Σέμνεμπι. Κύριο Στάλερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Πρέσβης. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε. θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι η κοινωνία της Γεωργίας από πολιτικής πλευράς είναι μια κοινωνία βαθιά πολλωμένη. Αυτή είναι η εντύπωση που είχαμε και σε επισκέψεις που είχαμε εκεί αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό που προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία μιας πολιτικής νοοτροπίας ενσωμάτωσης, ένταξης και όχι αποκλεισμού. Αυτό ήταν το καθήκον της αντιπροσωπείας που πήγε επί τόπου. Και αυτές οι ψευδείς ειδήσει στις οποίες συναφερθήκαμε πολλές φορές σήμερα, αποτελούν ένα παράδειγμα του αντίθετου, αν θέλετε, φαινομένου. Δηλαδή είναι μια πράξη αποκλεισμού ουσιαστικά από πολιτικής πλευράς. Συζητήσαμε με τον πρόεδρο και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μας είπε ότι το ντοκιμαντέρ αυτό ήταν, αν θέλετε, πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε πράγματι να είχε συμβεί. Πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι το ντοκιμαντέρ αυτό το οποίο ήταν σε θέση να πειράσει πολύ την κοινή γνώμη δεν προετοιμάστηκε εντελώ κατά τύχη. Δεν ήταν τυχαίο. Τώρα το ζήτημα των εκλογών και αν τελικά θα είναι αποτελεσματικές και αν τελικά θα λάβουν χώρα και στην Νότια Οσετία και την Αμπχασία, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε ραγλιστικά κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί δεν προβλέπεται επιτόπι δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Με αυτό συνδέεται και το ερώτημα της κυρίας Λόζινγκ για την ε, λεγόμενη νέα διεθνή ειρηνευτική δύναμη. Πρόκειται όντως ε, για μια δήλωση που γίνεται στις ε, συστάσεις του, που ενδεχομένω λάβατε και μέσω email. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αποστολή επιτήρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο βασικός παράγοντας σταθεροποίησης επιτόπου και όπως είπε ο κύριος Μορέλ θα πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσουμε την ε, ομάδα αυτή, την αντιπροσωπεία αυτή που κάνει μια καταπληκτική δουλειά και έχουν την πλήρη υποστήριξή μας. Το πρόβλημα είναι ότι ε, εξαιτία της ε, αρνητικής στάσης τόσο της Ρωσίας όσο και των επικεφαλής των περιοχών της Νότιας Οσετίας και της Απχασίας δεν είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περιοχές αυτές και γι' αυτό το λόγο υπόθηκε ότι θα ήταν καλό να υπήρχε μια διεθνής δύναμη η οποία να μπορεί να λειτουργεί και στις δύο πλευρές της διοικητικής διαχωριστικής γραμμής. Και αυτό άλλωστε έρχεται και η γεωργιανή πλευρά. Ολοκληρώνω λοιπόν στο σημείο αυτό. Είναι σαφές ότι ε, η θέση της Γεωργίας και η δική μας θέση είναι να έρθουν αυτοί και να τους φέρουμε κι εμείς πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα τελικό στόχο την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι ήδη έχουν γίνει κάποια πρώτα μέτρα όπως οι συμφωνίες α, σύνδεσης ή το νέο καθεστώς για την διευκόλυνση παροχής θεωρήσεων. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τάλερ για την παρουσίαση αυτή που μας κάνατε. Να ευχαριστήσω και τον πρέσβη Σέμνεμπη για την πολύ σημαντική συμβολή στην συζήτηση που έλαβε χώρα και να σε ευχαριστήσω όλους όσοι πήρατε το λόγο για να εκφράσετε τις απόψεις σας και για όσους έθεσαν ερωτήσεις. Α περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με την έκθεση του συναδέλφου Πεγιών για την Ένωση για τη Μεσόγειο. θα μας μιλήσει για τις πολλές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, καθώς επίσης και για τις συμβαστικές τροπολογίες στις οποίες έχει καταλήξει σε απόλυτο στονισμό με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου, προκειμένου να καταφέρει να μειώσει τον μεγάλο αριθμό των τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια του Μαΐου και θα την ψηφίσουμε την έκθεση στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Όσον αφορά τώρα τη Σύνοδο Ολομελίας, πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση για την έκθεση αυτή θα λάβει χώρα λίγες μέρες πριν την Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στις 7 Ιουνίου. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Μεσόγειος αποτελεί πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα της στρατηγικής μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα αυτό και μετά την εξέταση και έγκριση της έκθεσης αυτής. Προτού δώσω λοιπόν το λόγο στον συνάδελφο Πεγιόν, θα ήθελα να πω προς τους συναδέλφους ότι ακριβώς επειδή το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ζήτησα από τον κύριο Μεσαντέκ, τον Γενικό Γραμματέα για την Ευρώπη για τη Μεσόγειο, να συμμετέχει στην ε, συνεδρίασή μας πρόκειται να έρθει η συνεδρίαση που θα γίνει στις 23 Ιουνίου, δηλαδή αμέσως μετά την Σύνοδο Κορυφής της Βαρκελόνης. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έχουμε τότε την δυνατότητα να συζητήσουμε τα αποτελέσματα Τη ε, σημαντική αυτή συνόδου που θα λάβει η χώρα στη Βαρκελόνη μαζί με τον Γενικό Γραμματέα. Συνάδελφε Πεγιό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ιδιαίτερως ευχαριστώ για τα γενικά σας λόγια και την αποφασιστικότητα που δείξατε τώρα, εκφράζοντας την σημασία που έχει για την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο, το Σύμβουλο των Σχέσεων με τον Νότο και ιδιαίτερα η Ένωση για τη Μεσόγειο. Δεν θα ακρηγορήσω. Πάνω απ' όλα χρειάζεται εν ώψη τη αυριανή ψηφοφορία να ακούσω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να του ευχαριστήσω. Είχαμε θελήσει και ξέρουμε ότι δεν θα είναι απλό, θα χρειαστεί πολύ προσπάθεια και μονή να ε, προχωρήσει η Ένωση για τη Μεσόγειο. Χρειάζεται λοιπόν και αιμονή και επιμονή στη διαδικασία αυτή. Είχαμε πολλές τροπολογίες, 200, οι 60 κατά σημαντικό βαθμό, 90% ε, θα έλεγα, εμπλούτηναν το αρχικό κείμενο. και κατέστησαν πιο σαφή την διατύπωσή του και άρα ευχαριστώ τους και ηγητές από τις άλλες ε, πολιτικές ομάδες. Την κυρία Γιαννάκου με την οποία ακόμη σήμερα μιλήσαμε, την κυρία Γέγκλ, την κυρία Φλότχο. Γιατί από τις 25 συμβαστικές τροπολογίες που σας προτείνουμε, καταφέραμε πιστεύω κάθε φορά να λάβουμε υπόψη και τις ευαισθησίες ε, των μεν και των δε, και να εκφράσουμε ιδιαίτερες ευαισθησίες και προσδοκίες και ταυτόχρονα να ε, εκφράσουμε με σαφήνεια τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα ευχαριστώ τους κυρίους Κοπιόλς, ε, Κοπά, Μποντής, συναδέλφους οι οποίοι ιδιαίτερα ενεπλάξαν στην προσπάθεια αυτή. και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, βέβαια θα προκύψει και από τη συζήτηση, αλλά το βλέπουμε σαν αποτέλεσμα της λογικής μας ε, δουλειάς. Ένα θέμα θα ήθελα ιδιαίτερα να θίξω που με ανησυχεί και σας ανησυχεί όλους, από ό,τι γνωρίζω. Την έκθεση, όπως το υπενθυμίσετε και εσείς κύριε Πρόεδρε, επιλέξαμε να την αναπτύξουμε σε μια χρονική στιγμή που εξυπηρετεί και το στόχο της ε, πρόσδοσης μιας όθησης ε, να ενθαρρύνει δηλαδή τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων τον Ιούνιο γιατί κάτι δεν θέλει βέβαια να δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι δύσκολη η διαδικασία τη για τη Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προσκόμματα και έτσι θέλουμε το Κοινοβούλιο και να αδράξει την υπόθεση αυτή αλλά και να εκδηλώσει τις θέσεις του, την πολιτική του προτίμηση για μας, για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι σημαντικό όχι μόνο η επιτυχία, αλλά τα μέσα με τα οποία θα επιτύχει η, Ένωση για τη Μεσόγειο να προέρχονται από εμά. Και έτσι και πρέπει να σα πω ότι η Ιωνή για τον Ιούνιο, για τη μεγάλη αυτή σύνοδο του Ιουνίου, δεν είναι καλή. Κινδυνεύουμε ήδη από το Μάιο, δηλαδή από τη στιγμή κατά την οποία ψηφίζει το Κοινοβούλιο στην ολομέλειά του την έκθεση, να έχουμε εικόνα πολύ διαφορετική από ό,τι θα περιμέναμε ή θα επιθυμούσαμε. Και γι' αυτό θα, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ξανασυζητήσουμε σε ε, βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για να δούμε τι, τι στάση θα πρέπει να τηρήσει το Κοινοβούλιο εν προκειμένου μέσα σε ένα ε, κλίμα ίσως και κρίσης, ένα κλίμα πάντως δύσκολο. Περιεχόμενο. Ένα από τα πιο ακαθόδη ζητήματα ήταν βεβαίως τα άνθρωπα δικαιώματα και η θέση τους ιδιαίτερα η ισότητα ανδρών και γυναικών, ο πολιτισμός, ο διαπολιτισμικός διάλογος και διαθρησκιακός διάλογος, τα θέματα της ε, βιώσιμης φόρου ανάπτυξης και η λεπτή διαλεκτική μεταξύ της αναγκαιότητας να προχωρήσουμε μεταξύ ε, να προχωρήσουν συγκεκριμένα ε, σχέδια και εγχειρήματα που θα οδηγήσουν σε απεμπλοκή την κατάσταση στην Εγγύη και Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε προκειμένου να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο να βρούμε λύσεις ε, ορθολογικές πολιτικού ορθολογισμού που βρήκαν και βίκο αότα μερικές φορές συμπεριλαμβανομένες μάλιστα και της ενεργεία προεδρίας, ενώ αντίθετα υπάρχουν κάποιες τάσεις που οδηγούσαν σε ακόμη περισσότερες εμπλοκές και δυσκολίες. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους αναξαιρέτως τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Ένα-δύο θέματα μπορεί να έχουν μείνει που να χρήζουν ακόμη ε, επεξεργασίας. Υπάρχουν θέματα φερρυπίν της μετανάστευσης, το λεπτό αυτό θέμα στο οποίο πιστεύω έχουμε εξεύρει ικανοποιητική για τους μεν και τους δε συμβιβαστική λύση. Εάν όμως μένουν κάποιες εκκρεμότητες, πολύ ευχαρίστως να τις συζητήσουμε για να εκφράσουμε σαφή και περίφραστη θέση ως Κοινοβούλιο. Αυτή ήταν η δική μας τουλάχιστον φιλοδοξία. Η διαδικασία είναι ακαθόδης, είναι δύσκολη και πρέπει το Κοινοβούλιο να μιλήσει με σαφή και δυνατή φωνή. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Δίνω το λόγο στην κυρία Γιαννάκου, και ο για τρία λεπτά. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή, κύριο Πεγιόν, ε, για την ε, νομίζω πολύ σωστή κατεύθυνση εργασία που πραγματοποίησε για ένα ζήτημα που θα απασχολήσει φυσικά το Συμβούλιο γιατί είναι κατάλληλη στιγμή να στείλουμε ως Κοινοβούλιο ένα μήνυμα στο Συμβούλιο και βέβαια λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα πορεία της διαδικασίας της Βαρκελόνης. Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία της Βαρκελόνης μέχρι σήμερα δεν ικανοποίησε σε σχέση με τις φιλοδοξίες που είχαν αναπτυχθεί τότε. Πολλά προγράμματα παρέμειναν ε, ανεκμετάλλευτα και ανεκτέλεστα. Βεβαίως γίνεται αντιληπτό ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν διευκόλυνε ε, τη συνολική εξέλιξη αυτής της προσπάθειας. Ωστόσο, ε, η πρώτη αυτή προσέγγιση, δηλαδή η εμφάνιση δύο αξιωματούχων Ισραηλινού και Παλαιστινίου στη Γραμματεία, μας δίνει την ελπίδα όχι να λύσουμε εμείς το Μεσανατολικό, γιατί η Ευρώπη χρειάζεται πολλά βήματα ακόμη για να ρυθμίσει τέτοια ζητήματα, αλλά πάντως με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε ελπίδες, αλλά κυρίως Πρώτον για να μην υπάρξουν προσκόμματα στη γενικότερη προσπάθεια η οποία θα γίνει και δεύτερον γιατί ακόμα και κάτω από δυσμενείς συνθήκες πάντοτε υπάρχουν δυνατότητες <coughs> για να κάνει κανείς πολλά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, η συνεργασία, ε, η Ένωση για τη Μεσόγειο και η συνεργασία των μεσογειακών χωρών πράγματι δεν μπορεί παρά να εκταθεί σε όλους τους τομείς είναι σημαντικό το γεγονός ότι ενώ η Ευρώπη έχει χάσει πάρα πολλά από τα πολιτιστικά της ερίσματα και τους συμβολισμούς που την περιβάλλουν σε σχέση με το πώς τη βλέπουν οι χώρες στη Βόρεια Αφρική, ε, ωστόσο από την άλλη πλευρά δεν έχουν χαθεί όλα. Πιστεύω ότι υπάρχει διάθεση από όλες τις πλευρές ώστε η συνεργασία αυτή να επεκταθεί στην αηφόρο ανάπτυξη, στον πολιτισμό, στα θέματα παιδείας, φυσικά στα ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων και ισότητας των δύο φύλων και στις προσπάθειες που πρέπει και μπορούν να καταβάλουν αυτές οι χώρες για να επεκταθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς κανείς βεβαίως να θέλει να μη σεβαστεί την παράδοσή τους ε, και βέβαια σε ζητήματα προγραμμάτων που μπορούν να ωφελήσουν άμεσα τους ανθρώπους αυτούς και όλον αυτόν τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τα ζητήματα μετανάστευσης. Ε, γιατί η στήριξη των χωρών αυτών μπορεί να αποτρέψει σε κάποιο βαθμό ε, μια παράνομη μετανάστευση. Εκείνο που θέλω να σημειώσω κύριε Πρόεδρε είναι ότι σε μια τροπολογία που έχω καταθέσει εγώ την υπαριθμόν 39 υπάρχει σε ένα σημείο η φράση point of reference. Point de référence. Αυτό θα παρακαλούσα να διαγραφεί. Le point de référence. Ε, τελικά κύριε Πρόεδρε και συνολικά έχω την εντύπωση ότι η έκθεση με τις τροπολογίες έχει πράγματι εμπλουτιστεί και με τις τροπολογίες τις συμβιβαστικές Νομίζω ότι θα μπορέσουμε μέσω αυτού του εμπλουτισμού που κάνουμε στην έκθεση του συναδέλφου να δώσουμε μια ευρύτερη πολιτική διάσταση στη δουλειά που κάνουμε εδώ αλλά και ένα καθαρός πολιτικό μήνυμα για το πώς βλέπουμε την Ένωση για τη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γιαννάκου. Κυρία Φλότρα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εκεί που φτάσαμε στην επεξεργασία της έκθεσης και του συμβιβασμούς θέλω να ευχαριστήσω πρώτον ε, τον εισηγητή για, ε, για την προσπάθεια που κατέβαλε για να κατανοήσει όλα τα προβλήματα των συναδέλφων και φτάνουμε, καταλήξαμε μάλλον σε συμβιβασμούς που είναι ιδιαίτερα ισορροπημένοι. Ξέρετε πολλές φορές ε, οι συμβιβασμοί οδηγούν στο να μην λέμε πολλά πράγματα ενώ εδώ έχουμε συμβιβασμούς ε, πραγματικά με υπόσταση και καταφέρνουμε να συνδυάσουμε τις ανησυχίες και τον με και τον ε, δε. Υπάρχουν όμως μερικά προβλήματα ε, με τους συμβιβασμούς για τους οποίους η αμοιβαία θέληση του να καταλήξουμε κάπου δεν οδήγησαν στα προεξοφλημένα αποτελέσματα. <coughs> να σταθώ στις ε, δυσκολίες μας στον συμβιβασμό 11 σχετικά με τη Γεωργία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει συνένεση και πλειοψηφία για να υποστηρίξουμε τις διαπραγματεύσεις στην ΠΟΕ για τα γεωργικά ζητήματα. Αυτό όμως δεν αποτελεί και την πλειοψηφία της δικής μου πολιτικής ομάδας. Και ο συμβιβασμός 11 θα μπορούσε να υποστηριχθεί από την ομάδα μου στο βαθμό που θα αποφεύγαμε την αναφορά στις διαπραγματεύσεις της ΠΟΕ και να επιμείνουμε παραπάνω στην ε, ποιότητα της ε, γεωργικής πολιτικής ε, που θα στοχεύει στην τροφιμική ασφάλεια ή καλύτερα στην τροφιμική κυριαρχία. Πράγμα που θα θέλανε πολλά μέλη της ομάδας μου. Ο συμβιβασμός 13 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτός ο συμβιβασμός 13 πρέπει να είναι απόλυτα σαφής για το τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, ναι, να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως τις ηλιακές πηγές, απαντώντας στις ενεργειακές ανάγκες των χωρών της ε, Νοτίου Μεσογείου. Η αναφορά λοιπόν για μας να είναι υποδομές δικτύων νότου-νότου ε, και ρωτώ τον εισηγητή αν μπορεί να υποστηρίξει αυτή την παράγραφο, να γίνει δηλαδή σαφέστερα, σαφέστερη από ό,τι είναι, αναφερόμενος στις προκλήσεις στην νότια όχθη και να λυθούν τα ζητήματα του συμβιβασμού 11 επίσης. Πρέπει να πω ότι υποστηρίζω το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στις δύο όχθες και τα θέματα δικαιωμάτων ασύλου που για μένα είναι σημαντικότατα. Και να ολοκληρώνουμε με το συμβιβασμό 1. Εμείς έχουμε προηγούμενες ε, διατυπώσεις ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αυτή η αναφορά νομίζω στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εύστοχη και αν συμφωνεί ο εισηγητής θα μπορούσαμε να, να βάλουμε αυτή την αναφορά στο συμβιβασμό αριθμός 1. Ευχαριστώ κύριε Φλότρα. Ο συνάδελφος Μέγερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πεγιό ε, παρότι του, ότι η ομάδα μου παρουσίασε 40 τροπολογίες και καμία δεν συμπεριλήφθηκε στο συμβιβασμό. Εγώ αναγνωρίζω την προσπάθεια του κυρίου Πεγιόν για μία ε, σύνταξη που επιτρέπει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Εμείς ε, στις τροπολογίες μας θε, λέγαμε ότι οι μη λιμένες ε, συγκρούσεις αποτελούν εμπόδιο για την Μεσογειακή Ένωση και μιλάγαμε εδώ πιο συγκεκριμένα για την Παλαιστίνη. Ε, βέβαια είναι πολύ σημαντικό και η αναφορά που γίνεται για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, αλλά ξεχνιόνται και άλλα πράγματα, όπως είναι η Δυτική Σαχάρα, που βρίσκεται στα χέρια του ΟΓΕ και, είναι, και επίσης είναι και το θέμα της Βορείου Κύπρου. Η Κύπρος είναι χώρα της Ένωσης και εμείς καταθέσαμε μία τροπολογία όπου λέμε ότι η Τουρκία πρέπει να σέβεται όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Και η παρουσία 40.000 ε, στρατιωτών την Βόρεια Κύπρο δεν μας βοηθάει ε, στο να προχωρήσουμε σε μια πραγματική Ευρωπαϊκή ε, ε, Μεσογειακή Ένωση. Καταθέσαμε λοιπόν τροπολογίες αναφέροντας ποιες είναι εκείνες οι συγκρούσεις οι οποίες εμποδίζουν τη δημιουργία μιας Μεσογειακής Ένωσης. Τώρα διαπιστώσαμε με ικανοποίηση για, ε, μιλήσαμε για, την, για το ελεύθερο εμπόριο το οποίο ε, θα πρέπει να λαμβάνει όμως υπόψη του και την ασυμμετρία. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι με την αναφορά στο ελεύθερο εμπόριο αλλά δεν μας αρέσει το ότι αγνοείται η ασυμμετρία. Επίσης ε, δεν δεν συμφωνούμε με την ιδιωτική χρηματοδότηση, διότι εδώ αντιμετωπίζεται ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση, αλλά ε, θα θέλαμε και θα θέλαμε μάλλον να βρεθεί μία διατύπωση που να αποφεύγει αυτές τις ε, ε, προβληματικές για μας διατυπώσεις και αν, γίνουν αυτές οι διορθώσεις θα μπορούσαμε να ξαναδούμε τη στάση μας παρότι καταθέσαμε 40 τροπολογίες και δεν δεχθήκατε κανένα. Και πρέπει να επιμείνουμε στην σύγκρουση των συγκρούσεων που είναι το Παλαιστινιακό. Πρέπει να δοθεί ε, ένα, μετά, ένα ισχυρό μήνυμα αυτού του Κοινοβουλίου ότι πρέπει να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Μέγερ. Λόγω ο κύριος Γκέρενς, ο οποίος αντικαθιστά τον, τον σκιώδη συγητή της Άλντε, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως αντικαθιστώ τον σκιώδη συγητή. Δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στα αγγλικά και δεν μιλάω συνήθως στα αγγλικά. Εκπροσωπώ, όπως σας είπα, τον κύριο Βάγγεν, πολύ ταπεινά. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, αυτό είπαν και οι προλαλήσαντες. Η ομάδα Άλντε πιστεύει ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η εργασία που έχει γίνει για τις βασικές προτεραιότητες, μεταφορά, α, εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι προτεραιότητες αυτές για τις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες της Νότιας Όχθης, της Μεσογείου. Παρ' όλα αυτά απέχουμε πάρα πολύ από την εκπλήρωση των φιλοδοξιών μας και από τις ε, οι που γίνονται σήμερα έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Με ευχαρίστηση βλέπω ότι η γραμματεία στην Βαρκελόνη ε, αρχίζει και λειτουργεί πλήρως. Θα χρειαστεί όμως περισσότερος χρόνος ακόμα. Ήταν πολύ σημαντικό πάντως να διοριστεί γενικός γραμματέας και να αποφασίσουμε για το καταστατικό. Θα πρέπει τώρα να εξασφαλίσουμε ότι ε, η γραμματεία έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση και το απαραίτητο προσωπικό. Η προστιθέμενη αξία της Ένωσης για τη Μεσόγειο είναι ότι μπορεί να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό μας απομακρύνει από τις γενικόλογες μεγάλες πολιτικές συζητήσεις και εξασφαλίζει ότι από κοινού μπορούμε να λάβουμε την πραγματοποίηση πρακτικών προγραμμάτων όπως τα ενεργειακά προγράμματα τα οποία μπορούμε να έχουμε στη Μεσόγειο, ότι μπορούμε να προωθήσουμε την ανώτερη εκπαίδευση και τη συνεργασία σε πολλούς άλλους τομείς. Δεν μπορούμε όμως να αγνοούμε πως έχει κατάσταση στην, πραγματικό, στην, επιτόπου. Η α, κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να Τραβήξτε την προσοχή μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και οι δύο πλευρές στην ε, διένεξη στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για την εφαρμογή προγραμμάτων της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης. Επίσης, δεν θα πρέπει να διστάζουμε να ξεκινάμε ένα πολιτικό διάλογο με τους εταίρους μας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Μεσόγειος θα πρέπει να γίνει μια ζώνη ανοχής και ειρηνικής ε, συμβίωσης, συνύπαρξης διαφορετικών ε, πολιτισμών με διαφορετικές πεπιθήσεις. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μια στενότερη και πιο στενή, στενή με συνεργασία με τις χώρες της Νοτίου όχθης. Όντως υπάρχουν εδώ πέρα πάρα πολλές ευκαιρίες που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Θέλουμε περισσότερες επιχειρηματικές επενδύσεις, περισσότερη περιφερειακή ολοκλήρωση την πραγματοποίηση μεγαλύτερων project, σχεδίων. Χρειάζονται όμως τη βοήθειά μας οι εταίροι μας από την Νότια Όχθη προκειμένου να φέρουν εις πέρα σε όλα αυτά. Το ζήτημα της χρηματοδότησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να στεφθεί με επιτυχία η Ένωση για τη Μεσόγειο και τα επιμέρους προγράμματά της θα πρέπει να δώσουμε τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να διδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και το έχει ήδη κάνει. Έχει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα που θα επιτρέψουν τον συντονισμό κοινών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει ακόμα περισσότερο, να γίνουν περισσότερες επενδύσεις μέσω της ε, Euromed. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε την ε, δυνατότητα συμμετοχής ε, ιδιωτών επενδυτών στα project αυτά και να είμαστε προσεκτικοί βέβαια προς τη συμβολή τους. Θα Πρέπει επίσης ε, να τονίσουμε ποια είναι η στάση μας σε σχέση με τη συμβαστική τροπολογία 11. Πολλές φορές βλέπουμε ότι ε, Πρέπει να διατηρηθεί μάλλον η υπάρχουσα ορολογία και να μην χρησιμοποιήσουμε τη νέα ορολογία που προβλέπεται στην τροπολογία αυτή. Ευχαριστώ κύριε Γκέρενς, κυρία Κοπά και μετά ο κύριος Σομπιόλ και ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Δύο λεπτό καθένας. Κυρία Κοπά. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πεγιόν για τη δουλειά του, αλλά και την ικανότητα σύνθεσης που επέδειξε στις συμβιβαστικές του προτάσεις. Ήθελα επίσης να παρατηρήσω πως το μεγαλύτερο ποσοστό των προτινόμενων τροπολογιών των συναδέλφων τονίζει εμφατικά ότι χρειαζόμαστε τη συνεργασία στη Μεσόγειο. Επίσης, ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο δεν αντικαθιστά σε κανένα τρόπο, με κανένα τρόπο τη διαδικασία της Βαρκελόνης, αλλά αντίθετα χτίζει πάνω στο κεκτημένο της με σκοπό την αναθέρμανση της συνεργασίας μέσα από συγκεκριμένα κοινά προγράμματα. Αυτό που επιδιώκουμε πάντα είναι μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, μέσα από την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν ο πολιτικός διάλογος δεν χάνει τη σημασία του, αλλά ενισχύεται μέσα από τις επαφές σε κάθε επίπεδο, σε επίπεδο ηγετών, υπουργών, ειδικών, αλλά και σε αυτό το επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Συμφωνήσαμε όλοι ότι δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διένεξη και ότι δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην ανάγκη να υπάρξει επιτέλους λύση σε αυτό το πρόβλημα, όπως ευελπιστούμε να υπάρξει τελικά λύση και στο κυπριακό πρόβλημα, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις των τελευταίων ημέρων. Αυτό που προέχει εδώ όμως είναι να τονίσουμε ότι η δική μας άποψη είναι ότι η συνεργασία στους σημαντικούς τομείς χαμηλής πολιτικής όπως λέγονται, της Ένωσης για τη Μεσόγειο, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία και την εδραίωση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές. Εμπιστοσύνη που είναι αναγκαία όχι μόνο για την επίτευξη αλλά και βιωσιμότητα της μελλοντική λύσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των γυναικών, όπου θέλω να πω ότι θεωρώ εξαιρετικό το συμβιβασμό που επιτέχθηκε, καθώς και εδώ πιστεύω πως πρέπει να περάσουμε πια από τα ωραία λόγια στις πράξεις και κατά συνέπεια πρέπει πια να έχουμε ένα πρόγραμμα ειδικά για τις γυναίκες στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Ευχαριστώντας και πάλι τον ε, εισηγητή, ε, κλείνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κοπά. Δύο λεπτά για τον κύριο Μπιόλς. Πολύ σύντομα. Πρόκειται για μια καλή έκθεση. που αφορά ένα ζήτημα το οποίο δεν, είναι, δεν βρίσκεται σε μια ικανοποιητική κατάσταση. Εμείς θέλουμε η Ένωση για την Μεσόγειο να προχωρήσει, να θριαμβεύσει, να, έχει, να πετύχει αποτελέσματα να αντιμετωπίσει θετικά ε, αλλά η κρίση υπάρχει, υπάρχει ένα πρόβλημα ε, σχεδίου το οποίο θέλει πολιτικοποίηση μένα αλλά διαμορφώνει αυστηρά πολιτικά όργανα. Οπότε έχουμε μια παράλυση ε, λόγω του Μεσανατολικού στην Ένωση, την, στο προχώρημα της Ένωσης αυτής. Είδατε τι έγινε με τη διάσκεψη για το νερό που έγινε πριν από μερικές μέρες. Ο άλλος παράγοντας Πέρα δηλαδή από την ε, διαβρωτική ε, ε, διαβρωτική επίπτωση της, του Ισραηλοπαλαιστινιακού ζητήματος στην Ένωση για την Μεσόγειο λειτουργεί εξίσου διαβρωτικά και σε επίπεδο ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, δηλαδή με τη στάση που κρατάει ο καθένας αυτήν εδώ τη διένεξη. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους. Ευχαριστώ κύριο Μπιόλς. Ο κύριος Μποντής και η κυρία Βλαστό. Δύο λεπτά για τον κύριο Μποντής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Να συμφωνήσω με τους επένους για την έκθεση του κυρίου Πεγιόν, για το άνοιγμα πνεύματος που επέδειξε και για το πώς έλαβε υπόψη του όλες τις ε, προτάσεις τροπολογιών. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες ε, του συναδέλφου Πεγιόν και του συναδέλφου ε, ο Μπιόλ στην παραμονή της διάσκεψης του Ιουνίου Πρέπει λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο το Κοινοβούλιο να λάβει θέση και να ξαναπεί πόσο δεσμευμένο είναι στη διαδικασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Ήτανε πολύ επιτυχής η διάσκεψη κορυφής του Ιουλίου 2008, μας επέτρεψε να ξαναωθήσουμε την διαδικασία της Βαρκελόνης και είπαμε να μην περιμένουμε ε, την ε, πολιτική λύση, δηλαδή την ειρευτική Συμφωνία, στην Ισραηλοαραβική Διένευξη, αλλά να κοιτάξουμε να εργαστούμε ε, από κοινού για θέματα πολιτικής προστασίας, νερού κλπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όπως ε, ως θέση και ε, για το τουρκοκυπριακό και για ε, το πρόβλημα της Μαυριτανίας. Όμως νομίζω ότι για την... για το, για το Παλαιστινιακό Ισραηλινό ε, πρόβλημα έχουμε φτάσει στα όρια. Οι βομβαρδισμοί στην ε, Γάζα, η συμμαχία Νατανιάχου Λίμπερμαν υποσκάπτουν την ε, Ένωση για την Μεσόγειο. Δεν μπορούμε εμείς να ικανοποιηθούμε με, έναν, με μια κατανομή ρόλων όπου τελικά οι ΙΠΑ είναι αυτές οι οποίες αναζητούν την πολιτική λύση και η Ευρώπη πρέπει να ξεμπλέξει με θέματα χρηματοδότησης, καλής γειτονίας κλπ θα πρέπει τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Κομισιόν και το Συμβούλιο στα πλαίσια αυτής της συζήτησης να θυμίσουν αυτή τη λύση των δύο κρατών με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο. Ευχαριστώ. Η κυρία Βλαστό για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Καλό είναι η έκθεση αυτή για την Ένωση για τη Μεσόγειο να βρεθεί στο επίκεντρο των εργασιών μας, διότι θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαμορφώσει μια σαφή θέση πριν την συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο της Βαρκελόνης τον Ιούνιο. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση, γι' αυτό και μαζί με τους συναδέλφους Σαϊφή, Μποντής και Φράνκο ε, θεωρήσαμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε μια σειρά από πολιτικές προτεραιότητες, δηλαδή ασφάλεια της πρόσβασης στην ενέργεια, ε, εκκίνηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να ξεκινήσει η ανάκαμψη οικονομίας και να προσελκύσουμε τους επενδυτές. Η εναντήρια εκπαίδευση, η έρευνα, η επιστήμη, ένα ευρωμεσογειακό ενδεχομένω Ινστιτούτο των ε, διερεύνησης των δασικών πυρκαγιών. Είναι διάφορα σχέδια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την οικονομική και εμπορική ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών του Νότου και όχι μόνο να αναπτύξουμε σχέσεις βορρά-νότου. Θέλουμε διμερείς σχέσεις. Η δε περιφερειακή ολοκλήρωση του Νότου αποτελεί όρο κτηνών κάνευ για την επιτυχία αυτής της εταιρική σχέσης και θα πρέπει και η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση να συμβάλλει. Μαζί με τον κύριο Πεγιόν, λοιπόν, μπορέσαμε να βρούμε ικανοποιητικέ για μας συμβαστικές λύσεις. Τον ευχαριστώ. Η διαβούλευση μας επιτρέπει σήμερα να έχουμε μπροστά μας ένα σχέδιο έκθεσης ολοκληρωμένο, ισορροπημένο, γερό, ένα σχέδιο το οποίο θα υποστηρίξουν ευρύτατα πιστεύω οι συνάδελφοι και το οποίο ελπίζω θα ληφθεί υπόψη στη συνέχεια από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βλαστό. Ο κύριος Πενιό για την τελική απάντηση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Η παρατήρηση της κυρία Φλότρου νωρίτερα ήταν πολύ εύστοχη και από την κυρία Βλαστό επίση αποκόμισε το εντύ, την εντύπωση ότι δεν είναι απαραίτητα ορθός ο όρος συμβιβασμός για την κοινή μας δουλειά. Γιατί δεν νομίζω ότι προσπάθησε κανείς ή δέχτηκε κανείς να υπαναχωρήσει σχέση με τις θέσεις του. Απλώς προσπαθήσαμε να τις εμπλουτίνουμε περισσότερο και καταλήξαμε σε πολύ καλά αποτελέσματα. Ε, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Ε, μάλλον έχουν εμπλουτίνει το κείμενο οι διαφορές ε, ε, τροπολογίες χωρίς να οδηγήσουν σε συμβιβασμό. Δηλαδή ουσιαστικά συνεχίζουμε στην αρχική πορεία του κειμένου κάθε φορά. Αυτό είναι το πνεύμα που επικράτησε. Και δεύτερον, δεν θα ήθελα γιατί θα ήταν αντίθετο με την φιλοσοφία μας. Δεν θα ήθελα να δοθεί εντύπωση ότι η μόνη δυσκολία που αντιμετωπίζει η Ένωση για την Μεσόγειο είναι η Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Είναι ένας από τους παράγοντες, μία από τις δυσκολίε η Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση και άλλωστε το έχουμε λάβει υπόψη, το έχουμε σημειώσει και στην τελική μορφή του κειμένου με μία ε, τροπολογία βεβαίω όπου επιμένουμε να ε, αναγνωριστούν τα δύο κράτη με κοινή πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ κτλ. Την, την κοινή θέση δηλαδή, του Κοινοβουλίου, χωρίς όμως και να πρέπει να παρασυρθούμε στην εντύπωση ότι δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Η Κύπρος, η Δυτική Σαχάρα και πολλά άλλα, αγαπητέ κύριο Βιόλς. Αυτά που είδαμε το τελευταίο καιρό σχετικά με την Τουρκία, Φερρυπίν. Οι δυσκολίες δηλαδή που έχουμε με τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο και μετά τη Γάζα και μετά το αδιέξοδο που αντιμετωπίσαμε στην υπόθεση αυτή την Ισραηλοπλαιστινιακή σύγκρουση. Και πέραν αυτής όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, άλλες δυσκολίες. Για δε τις κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεγάλη δυσκολία. Γιατί? Γιατί είχαμε συνηθίσει με την πολιτική της ε, γειτονίας, με τις διμερείς σχέσεις, που ορισμένοι μάλιστα είχαν βολευτεί πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο όμως να πείσουμε τώρα τους εταίρους της Νότιας Όχθης ότι τώρα έχουμε άλλη πλέον δομή, έχουμε συναπόφαση, έχουμε συνυπευθυνότητα, έχουμε συνύπαρξη, περιφερειακή συνεργασία για την ακρίβεια. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην εξυπηρετήσουμε εκείνους, από το Ισραήλ ίσως, αλλά οπωσδήποτε και από την Παλαιστίνη, που τάσσονται κατά των εξελίξεων. Πάντω η έκθεση καταγράφει, υπενθυμίζει ξεκάθαρα τη θέση μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να την αποδεχθούμε όλοι. Γιατί δεν την Κύπρο. Προτάθηκαν τροπολογίε, Ακόμη και σήμερα το πρωί τι συζητήσαμε. Μέχρι αύριο το πρωί θα επιδιώξω να διατυπώσω μία διαπρόταση που να γίνεται δεκτή από τους πάντες, μία διατύπωση η οποία θα ήταν, θα έλεγα, λογική να μην οδηγεί δηλαδή σε περαιτέρω εμπλοκές και ταυτόχρονα υπενθυμίζει ποιες είναι οι αρχές μας. Στη συνάδελφα κυρία Φλότρο επεσήμανα ότι δεν έχω αντίρρηση ως προς το ζήτημα των συλλογικών δικαιωμάτων, άρα θα τα επανεισαγάγουμε στο κείμενο. Πρόβλημα ως προς την κατανόηση μόνο μπορεί να υπήρξε ε, για το τι εννοούσα εγώ ως δικαίωμα πρόσβαση στα δημόσια αγαθά θεωρούσα ότι ήταν ήδη αρκετά μακροσκελής ο κατάλογος που είχαμε στην πρώτη έκδοση. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και η σχέση με αυτόν, νομίζω ότι στο θέμα αυτό, από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρξει πλειοψηφία με τη στάση που τηρεί και η δική σας ομάδα, κυρία Φλότρο, προς την τήρηση των όρων του ΠΟΕ. Και για το τελευταίο σημείο, τα δίκτυα βορρά-νότου για την ενέργεια, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λειτουργήσει αμφίδρομα. Αλλά νομίζω ότι ξεκάθαρα είπαμε, και σας διαβάζω, στη συμβαστική υπαριθμό 13, ότι επιθυμεί τα σχέδια να αναπτύσσονται και κατά προτεραιότητα με γνώμονα τις ανάγκες των κρατών που τα ζητούν. Δηλαδή να αποβαίνουν σε όφελο των κρατών του Νότου, τη Νότια Όχθη, κατά προτεραιότητα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν και ανταλλαγέ, να μην αμφίδρομοι οι σχέσει μεταξύ Βορρά και Νότου. Θα ήταν παράλογο κάτι τέτοιο στην Ένωση για τη Μεσόγειο, αν το ζητούσαμε. Αυτά. Εάν μέχρι αύριο το πρωί μπορέσουμε είτε για την επιστηστική ασφάλεια, είτε για κάποια άλλα σημεία να βρούμε διατύπωση που να βελτιώνει το κείμενο πολύ ευχαρίστω. Εν γέννη πιστεύω διατυπώνονται σαφ σαφείς τοποθετήσει από πλευράς της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως και για την προφορική σας τροπολογία που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο στο στόχο της ε, συμβαστικής ε, τροπολογίας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και για, την, ε, για το προϊόν αυτό της κοινή μας ε, προσπάθειας, ε, το κείμενο αυτό το οποίο πιστεύω θα έρθει την κατάλληλη στιγμή στις πολιτικές ζυμώσεις και τη μεγάλη διάσκεψη για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή Πεγιών. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι όντω η δουλειά του ήταν καταπληκτική και δίνω την προεδρία στον κύριο Μποντής, ο οποίος θα ασχοληθεί και με το τελευταίο ζήτημα στη μερίσια διάταξη. Χαίρετε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 Euh, Θα εξετάσουμε τώρα την έκθεση που έχει να κάνει με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δίνω το λόγο στην κυρία Χαουτάλα για να μας παρουσιάσει τις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ως στόχο να κατευθύνει τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εδώ πέρα πιο ισχυροί μηχανισμοί και να υπάρχει μια πιο συστηματική προσέγγιση πλέον. Αυτή τη στιγμή συνθήκη τη Λισαβόνα ενισχύει τις υποχρώσεις που έχουμε για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης θελήσαμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο, καθώς επίσης και με διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται για την υπεράσπιση των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρομαι για παράδειγμα στα Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τέλος, ήταν πολύ σημαντικό το ότι ήρθαμε σε επαφή με οργανώσεις των πολιτών που υπερασπίζουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή αύριο και χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετείχαν πάρα πολύ στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής και πραγματικά ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα αντιπροσωπεύει πραγματικά την πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι με αυτή θα συμφωνήσουν και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνω ότι η ύπατη εκπρόσωπος είπε ότι θέλει να είναι παρούσα στην συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια τον Ιούνιο για την έκθεση αυτή. όπου θα συζητηθεί και η ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τόσες πολλές τροπολογίες. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι κανείς πάντα ικανοποιημένο για έναν τέτοιο μεγάλο αριθμό τροπολογιών, 170 στο σύνολό τους, αλλά αυτή τη φορά κατάλαβα ότι ουσιαστικά οι συνάδελφοι ήθελαν να βελτιώσουν το κείμενο. Επομένως, σχεδόν τα πάντα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να ενταχθούν στο βασικό κείμενο. Στον κατάλογο ψηφοφορίες βλέπετε τώρα μία σειρά συμβαστικών τροπολογιών που κατά την άποψή μου καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος τροπολογιών που υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Να αφαιρθώ σε δύο ιδιαίτερα ζητήματα. Στην τροπολογία 40, στόχος εδώ πέρα ήταν να έχουμε μια, έναν ενοποιημένο ορισμό όσον αφορά τον υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προτείνω να μην εγκριθεί η τροπολογία αυτή, αλλά να εγκριθεί η τροπολογία 28 η οποία αναφέρεται σε έναν ορισμό που περιλαμβάνεται και στη διακήρυξη των Εθνών για του υπερασπιστέ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1998. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποια αυταρχικά καθεστώτα τα οποία θα επιθυμούσαν έναν πιο στενό, περιορισμένο ορισμό των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακριβώ για να μην υπερασπιστούν τελικά του ανθρώπου αυτού. Γι' αυτό το λόγο σα ζητώ να υπερψηφίσετε την τροπολογία 28 αντί τη τροπολογία 40. Επίσης, χρειάστηκε να απορρίψω την τροπολογία 52 που αναφέρεται σε περιφερειακές και περιφερειακές θεματικές στρατηγικές όσον αφορά τους περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο σχέδιο έκθεσης στο συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου αναφέρεται στην πολύ μεγάλη σημασία των τοπικών στρατηγικών που εφαρμόζουν οι αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες υποστηρίζουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχω να προσθέσω άλλα πράγματα και ελπίζω ότι οι πολιτικές ομάδες έμειναν ικανοποιημένες από τις επραγματεύσεις που έλαβαν χώρα και που πιστεύω ότι αντικατοπτρίζονται και στην λίστα, στον κατάλογο ψηφοριών. Από δική μου πλευρά θα υπάρχουν και κάποιες προφορικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. ποιο επιθυμεί να πάρει το λόγο. Κύριε Γιαννάκου. Κύριε κύριε Ε, θέλω να σημειώσω, πραγματικά υπάρχουν ε, τροπολογίες συμβαστικές και θέλω να συγχαρώ την κυρία Χαουτάλα για την έκθεσή της. Αυτό που θέλω να σημειώσω σε σχέση με τροπολογία 40, επειδή πράγματι η δική σας τροπολογία, κυρία Χαουτάλα, 28, λέει εντελώς το αντίθετο από αυτό που λέω εγώ στην τροπολογία 40, δηλαδή ο όρος του Ηνωμένων Εθνών του 1998 πράγματι παραμένει πάρα πολύ ασαφής και εγώ θα ήθελα ίσως ένα πιο συγκεκριμένο ορισμό. Ε, προτείνω τον εξή συμβιβασμό που νομίζω ότι μπορεί να δεχτούμε την τροπολογία τη δική σας, την τροπολογία 28 και να προσθέσουμε αντί της δικής μου τροπολογίας την εξής φράση considers that the EU based on the United Nations Declaration of 98 should further θεωρεί ότι θα πρέπει περαιτέρω η δήλωση των ΗΕ να ε, αναπτύξει τα δικαιώματα των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά την δήλωση του 1998, έτσι ώστε να αξιολογείται καλύτερα η δουλειά του και να αναπτύσσεται προκειμένου να υπηρετούν καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει συνδυασμό ε, της 28 και τη 40, ε, χωρίς να έρχονται σε αντίθεση, σε αντίθεση μεταξύ τους, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Madame Vergia. Κυρία Βεργιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστώ την κυρία Χάουτολα για τις προτάσεις της και την κατάθεση των ε, τροπολογιών. Οι συμβαστικές τροπολογίες σε μεγάλο βαθμό καλύπτουν τις τροπολογίες της ε, ομάδας μας, της ε, Νοτικής Αριστεράς. Ένα πράγμα μόνο. Για ένα πράγμα μόνο λυπάμαι, ότι η κυρία Χάουταρα από ό,τι βλέπω συχνά υποτάσσεται πυθύνια στις αρχές, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ατίθασοι και πιο αποφασιστική στις, ε, στα αιτήματα που, ζητώ, που διατυπώνουμε. Και την ευχαριστώ βεβαίως για τις προτάσεις της. Για τις λεγόμενες κυρώσεις, εντός εισαγωγικών χρησιμοποιώ τον όρο, γιατί μάλλον αρκετά ε, είναι υπερβολικά ε, αυστηρός, αλλά κάποιου είδους κυρώσεις πρέπει να υπάρχουν για τις παραβάσεις και επίσης ένα ερωτηματικό για ένα σημείο πολύ μικρό, αλλά πάντως που με παραξενεύει πολύ. Στην τροπολογία 27, όπου ζητάτε σε χωριστή ψηφοφορία στο τέλος της ε, τροπολογίας, χωρίς να απορρίπτετε την πρότασή μου για την ασφάλεια των οικογενειών. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ξέρετε ότι πολύ συχνά τις οικογένειες των ε, αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις χρησιμοποιούν ε, για να τους ασκήσουν πιέσεις, να τους υποχρεώσουν να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους. Και εν πάση περιπτώσει, πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο γίνεται με τρόπο πιο αποφασιστικό και πιο απερίφραστο, να μην βλέπουμε συχνά και μέσα στο Κοινοβούλιο αλλά και σε επίπεδο Επιτροπής και Συμβουλίου να αντιτυπώνονται λόγια που δεν βρίσκουν το αντίστοιχό τους στις πράξεις. Θα ήθελα δεν να σημειώσω ότι ένα από τα πιο ικανοποιητικά παραδείγματα του τελευταίου καιρού ήταν ε, ε, αυτό που έχουμε δει σε σχέση με την Τινησία. Έχαμε διαρκείς εκκλήσεις ε, για την ε, κατάσταση στην Τινησία και είναι δυστύχημα θεωρώ το ότι έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την χώρα αυτή. Κύριε Χάουταλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Γιαννάκου. Τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση για το στόχο που προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε με την ε, τροπολογία αυτή της τελευταίας στιγμής. Αλλά θα ήθελα να πω ότι εάν ζητήσουμε, ε, να προαχθεί περισσότερο ορισμός, ε, να εξελιχθεί περισσότερο ορισμός των αγωνιστών κτλ. όπως προτείνεται, υπάρχει ο εξής κίνδυνος. ίσως ορισμένε χώρε και αυτή ίσω είναι και η τάση στο Συμβούλιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα, Συμβούλιο Ασφαλεία κτλ. να αποκλείσουν από την κατηγορία αυτή κάποιες, ε, αγωνιστές και ίσως να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο, δηλαδή του ορισμού ή του, της επέκτασης του ορισμού για τους στόχους τους. Και τι, όπως είπα, σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα το στόχο που προσπαθείτε να επιδιώξετε. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Για την κυρία Βιώνα. Ναι, για την τροπολογία 27. Οι οικογένειες και συγγενικά πρόσωπα έχουν προσθεθεί στο κείμενο, όπως ζητήσατε. Εγώ δεν θέλησα απλώς να χρησιμοποιήσω τον όρο άμυνα, γιατί είναι σκοπιμότερο να μπει ο όρος προστασία μέσα στο κείμενο. Σημειολογικό ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά πάντως ε, άτομα ε, και εκεί, ναι, τους έχω λάβει υπόψη, τους έχω συμπεριλάβει στο κείμενό μου και ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τη συνεργασία μέχρι αυτή τη τελική στιγμή του εγγράφου. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Για όποιον ενδιαφέρεται, επισημαίνω ότι το Προεδρείο, το Διευρυμένο Προεδρείο θα συνεδριάσει στις 6.30 σήμερα το βράδυ. Η Επιτροπή μας αύριο το πρωί κάνει τις ψηφοφορίες 10 και 30. Σας ευχαριστώ. Πέρα συνεδριάσεως.